So what we have now, we have only the first, uh, only this, or we have four at the same time, individually? Yeah, yeah, yeah. yeah. Individually, no, no, one by one. Uh, Report per report. That's, That's report. So in the discussion, okay. Uh, Dear colleagues, I would like to start the... Αγαπητοί συνάδελφοι, θα παρακαλούσα να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Η Κωνσταντς είναι εδώ. Είστε μακριά ένας από τον άλλον, θα είναι πολύ δύσκολο. Αλλά εν πάση είναι μικρή αίθουσα. Καλά. Ξεκινάμε λοιπόν με την εξέταση του σχεδίου εκθέσεως της Κωνσταντς ε, Κρέλε και του Λάμπερτ Φαν Κρέλε και του Λάμπερτ Φαν Νίστιλροι. Φαντάζομαι ότι θέλετε εσείς να κάνετε την παρουσίαση και την εισήγηση για την συζήτηση. Θέλετε να πείτε δύο λόγια, Κωνσταντς και Λάμπερτ. Σύντομα, σύντομα έτσι, να δώσετε και το καλό παράδειγμα εσείς. για να διατηρήσουμε και το καλό πνεύμα που είχαμε το πρωί, Πρόεδρε. Αφού ακούσαμε και τους ε, εκπροσώπους των ε, περιφερειακών ε, οργανώσεων, γενικών οργανώσεων, ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν προτάσεις και τροπολογίες και ιδέες που ταιριάζουν με την άλλη. Το μικρόφωνο του μιλητή έχει κλείσει, αλλά είναι ανοιχτό το μικρόφωνο της Προέδρου. Λοιπόν, και με το θέμα αν, είναι, αν υπάρχουν τροπολογίες, αν δεν υπάρχουν τροπολογίες. Είδαμε ότι περιμένουμε νέες τροπολογίες θα περάσουν από τη μετάφραση, θα βρούμε την κατάλληλη στιγμή για να τις ε, συστήσουμε και αυτές. Άρα έχουν πει τα πράγματα στο δρόμο τους. Οι παρατηρήσεις μου είναι δύο. για την ε, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, τα θέματα αυτά που συστήσαμε δηλαδή σήμερα. Έχουμε επισημάνει ότι μπορεί κάθε χώρα, μπορεί ή θα έπρεπε καλύτερα κάθε χώρα να θεσπίσει μια, εταιρεία συμφωνη... μια εταιρική σχέση, μια συμφωνία εταιρική σχέση, ένα εδαφικό σύμφωνο όπως θα το λέγαμε παλιά, που θα επιτρέπει να ενισχυθεί η επικουρικότητα και ο ρόλος των εταίρων χωρίς να επιβαρυνόμαστε με περισσότερη γραφειοκρατία. Και επί παραδείγματι, εάν το συμφωνοτερικής σχέση ε, αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή θα έχει εκείνη την ευκαιρία μέσα σε ένα τρίμηνο να το εξετάσει. Ίσως και οι εταίροι μέσα στο διάστημα αυτό θα μπορούν να το συμπληρώσουν και το καθεξής. Δηλαδή μια διαδικασία ευέλικτη, ανεκτή, να μην γίνονται και κλεισμένο των θυρών συστήσεις και να γίνονται αποφάσεις εν κρυπτό και παραβίστο. Και έτσι, για το άρθρο 46 προβλέπουμε μία πρόταση, μία ε, έκθεση προόδου που θα υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, για τις εξελίξεις στις ε, συμφωνίες αυτές, συμβάσεις αυτές. Επίσης, για το άρθρο 46 και 5 λέμε ότι θέλουμε να υπάρξει ο παραλυσμός ε, με την Ευρώπη του 2020. Η παράλληλη πορεία. Και όπως βλέπετε ε, προσπαθούμε να διευκρινίσουμε τις προτάσεις μας όπου αυτό χρειάζεται. Στην αιτιολογική σκέψη 15, τροπολογία 6, Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω εντωμεταξύ ότι πρόκειται να ε, καταθέσω προτάσεις συγκεκριμένες για προσέγγιση του ορίζοντα 2020 και το Ταμείο. Γιατί λέμε ότι στο Ταμείο περιφερειακή Ανάπτυξης ζητούμε, όπως λέει το άρθρο 60, από κάθε περιφέρεια να δαπανά τα κονδύλια σε συνεργασία με τις άλλες περιφέρειες. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή να συμμετέχει κανεί με συνεργασία, όχι μόνο σε επίπεδο ευρωπαϊκής εδαφικής αλλά και σαν στάση εθνική να συμμετέχουμε, να ε, συνεργαζόμαστε μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που μπορεί να αποτελέσει πιστεύω μια εξαιρετική, μια βασιλική οδό προς ε, την ε, αριστεία την οποία επιδιώκουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις περιφέρειες. Αυτά δεν ξέρω αν η Κωνσταντς έχει. Α, ναι, έχουμε και το ε, το κοινωνικό ταμείο, αν έχει, κάτι να συμπληρώσει. Ναι, Λάμπερτ, ευχαριστώ πολύ. Ίσως θα χρειαστεί να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες τροπολογίες που θα δείτε στο δεύτερο γύρο. Άρθρο 4 και 95, προγραμμάτα εθνικών μεταρρυθμίσεων, όπου προτείνουμε την χρήση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων ως βάση αναφοράς για τις συστάσεις ανά έτος, ε, διότι θεωρούμε ότι αυτά τα προγράμματα, τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης είναι μακροπρόθεσμα προγράμματα μεταρρύθμισης, ε, περιγράφουν τις εθνικές μεταρρυθμίσεις, υπογραμμίζουν την ανάγκη για ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα. Και δεδομένου ότι θεωρούμε ότι τα ελληνικά πρωτογράμματα σε ε, συμβαστερικής σχέσης αποτελούν ε, έναν, ε, μια εξέλιξη μακροπρόθεσμη. θέλουμε τέτοια προγράμματα να τα έχουμε μέσα στο έγγραφο. Ιδάλλως, θα είχαμε δύο διαφορετικά ήδη δύο διαφορετικές κατηγορίες εγγράφων με δύο διαφορετικές ταχύτητες. Αυτό ε, εξηγεί τις τροπολογίες. Το άλλο θέμα που θέλω να προτείνω θα ήταν και ίσως οι πιο παλιοί θυμούνται. Ο κύριος Χατζηδάκης από την προηγούμενη θητεία είχε καταθέσει τη σχετική πρόταση στον κανονισμό τελευταία φορά, προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες, ισότητα των φύλων, προκλήσεις σχετικές με την ισότητα των φύλων και σχετικές προκλήσεις. Θεωρούμε ότι αυτές οι κατηγορίες των γυναικών, των ατόμων με ειδικέ ανάγκες, των ατόμων που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας, ε, πρέπει να υπογραμμιστούν ιδιαίτερα στην ε, πολιτική και εδώ η γενίκευση της ε, εξάντα αιρεσιμότητας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ξέρουμε ότι η Προεδρία της Δανίας έχει προτείνει κάτι διαφορετικό, αλλά εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί αυτή η γενική οριζόντια αρχή στο γενικό κανονισμό και είναι πιστεύουμε πολύ σημαντικό να έχουμε και τον ε, γενικό κανονισμό και την ε, εκ των προτέρων αρισιμότητα. Για τις ε, τροπολογίες έχουμε ένα κατάλογο 7, 14, 48, 87, 101 και δύο είναι τα ε, νούμερα των άρθρων που τροποποιούνται με τις τροπολογίες μας στη δεύτερη αυτή φάση. Τα άλλα αφορούν νομίζω μόνο θέματα Και έχουμε τροπολογίες για, τις, ε, για τα δημοσιονομικά μέσα, οριζόντια πάλι ζητήματα όπου βλέπουμε ότι τα δημοσιονομικά μέσα είναι σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης, ε, μάλλον στον προγραμματισμό για τις περιφέρειες και θέλουμε να τηρήσουμε αυτή την ε, τάξη, αλλά χρειάζεται περισσότερη διευκρίνηση των κανόνων. Γι' αυτό ρωτήνουμε και τις σχετικές τροπολογίες. Φερρυπίν, στόχος δημοσιονομικών μέσων που λέει η Επιτροπή Νόρος που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν αναγνωρίζουμε πουθενά στο κείμενο του κανονισμού αυτόν τον όρο και γι' αυτό πρέπει να τον τροποποιήσουμε για να διευκρινίσουμε πώς ακριβώς μπορούν να είναι οι κανόνες που θα αναπτυχθούν στο μέλλον για τα δημοσιονομικά μέσα. Από την άλλη, με τις ε, τροπολογίες μας καθιστούμε σαφές ότι χρειαζόμαστε κάποιους βασικούς κανόνες ήδη από το Γενικό Κανονισμό και όχι μόνο στις ε, πράξη, Νομίζω ότι θα πρέπει να το σημειώνουμε στο Γενικό Κανονισμό. Χρειάζονται επίσης τροπολογίες για την τεχνολογική υποστήριξη. Ήδη είχαμε συζητήσει για την ενίσχυση τη ε, δυνατότητα των εταίρων, συμμετοχή στην εταιρική σχέση και τώρα στα άρθρα 51-52 επισημαίνουμε ότι δεν είναι απλώ απαραίτητο ή δυνατόν να αξιοποιείται η δυνατο να αξιοποιειται υποστήριξη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή από του εταίρου, αλλά θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να την αξιοποιούν και να προσφέρουν με την πλευρά από την πλευρά τους ανάπτυξη δυνατοτήτων. Άρα ένα σημαντικό θέμα αυτό. Και επίσης ερχόμαστε στο περίμενο CSF που θα ήθελα να σας εξηγήσω λίγο τι σημαίνει. Ε, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο λοιπόν θέλω να σα εξηγήσουμε το έχουμε συμπεριλάβει στο, στο παράρτημα για το γενικό κανονισμό και είπαμε την προηγούμενη φορά ότι θα καταθέταμε τροπολογία. Ήταν υπερβολικά ε, φιλόδοξη αυτή η πρόβλεψη. Τελικά λοιπόν έχουμε περιοριστεί σε ένα άτυπο έγγραφο εργασία για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο όπου προτείνουμε τη ραχοκοκαλιά του Κουσουπού την οποία θα πρέπει ναι, να συζητήσουμε και αν συμφωνείτε, γιατί είχαμε προετοιμάσει και άλλα πράγματα, αλλά θέλαμε να, να, περιοριστούμε μόνο σε μικρό όγκο για να μπορείτε να διαβάσετε αυτές τις δύο-δυόμιση σελίδες, να ε, δείτε τι αποσκοπούμε με αυτό το, το γενικό ρήφημα και να τοποθετηθείτε πάνω σε αυτό. Συντονισμός μεταξύ των ταμείων που οργανώνει ο Γενικός κανονισμό Γεωργία, Αλία, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ταμείο Συνοχής, ενσωματώνοντα αυτό και επίση ενσωματώνονται και Επισωματώνονται αυτά πάνω στι λοιπέ πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρει πριν το 2020, Κόσμο Life, ΚΥΠΑ, EDF, ε, Ευρωπαϊκό Τομέα Ανάπτυξη, Εράσμου για όλους και άλλα αντίστοιχα προγράμματα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειακών προγραμμάτων και των λοιπόν ευρωπαϊκών πολιτικών. Και αρνεστούμε βέβαια την καταλληλότερη διατύπωση δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο key action, κέρια δράση, αλλά ε, και αυτό γιατί δεν υπάρχει πουθενά αλλού, α, δεν υπάρχει ως ορισμός πουθενά, αλλά σκεφτόμαστε κάτι σαν κέριο στόχος και target, που θα μπορούσε να είναι μια χρήσιμη έννοια. Το βλέπετε και στο εγγραφείο εργασία. ότι προσπαθούμε να συνδυάσουμε τα μέσα των διαφόρων ταμείων και να τα ενσωματώσουμε στις προοπτικές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τηρώντας βέβαια και τις προϋποθέσεις των λοιπόν μέσων της ευρωπαϊκής ε, πολιτικής. Θα θέλαμε να επισημάνουμε τους στόχους οριοζόντιους αλλά και προκλήσεις συγκεκριμένες πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, βιώσιμη ανάπτυξη, συνεργα... Ε, ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, απαγόρευση διακρίσεων, προσβασιμότητα, ολοκληρωμένη προσέγγιση. Όλα αυτά είναι οι ιδέες που έχουμε να προτείνουμε. Ιδέες που θα θέλαμε να υλοποιήσουμε εξασφαλίζοντας βέβαια το περιεχόμενό τους όπως αυτό έπαιτε και υλοποιώντας τις, ή προχωρώντας της για υλοποίηση το έχετε δυνατό ίσως με, ένα, με την πρόβλεψη για κείμενο στην προσοχή μας Εδρία ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε στις 29 Μαΐου όπου, και προτείνουμε, όπου θα προτείνουμε μάλλον την διαδικασία. Γι' αυτό προτείνουμε σήμερα να έχουμε προτάσεις για τροπολογία μέχρι την 1η Ιουνίου. Για να παρακολουθήσουμε το κοινό στρατηγικό πλαίσιο στο δυνατόν πιο πιστά. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Και ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να την στηρίξει, να υποστηρίξει τις προτάσεις μας και να μας προσφέρει αρρωγή ώστε να βρούμε την καταλληλότερη διατύπωση για το παράρτημα. Μέχρι τώρα η Επιτροπή δεν φαινόταν έτοιμη να προσφέρει την υποστήριξη αυτή. Ιδάλλωστε είχαμε διατυπώσει την τροπολογία για ολόκληρο το περιεχόμενο, αλλά ίσως στη ε, συνάντησή μας τη σημερινή, ίσως σήμερα, στη συνεδρίαση αυτή να μπορούμε να δούμε κάποιες λύσεις για το παράρτημα ώστε να τις διατυπώσουμε πιο συγκεκριμένα και να ληφθεί η απόφαση μέχρι τον Ιούλιο στην Επιτροπή. Λυπούμε αν μακρηγόρησα, αλλά έπρεπε να γίνει αυτή η εισαγωγή. Ωραία. Προχωράμε στους κοιόδης Δεν βλέπω τον κύριο Γκουτμάνη αυτή τη στιγμή. Ελίζα Μπεσρέτερ. Απουσιάζει και εκείνη. Όλτζερ Βλάσακ ακόμα είναι παρόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ και να επενέσω τους ε, συναδέλφους συνεισηγητές. Νομίζω ότι πολλά είναι τα ζητήματα που ανακύπτουν εδώ και ε, περιλήφθηκαν όπως και οι παρατηρήσεις των περιφερειακών οργανώσεων. Αυτό δείχνει το πνεύμα συνεργασίας και την προθυμία και διαλεκτικότητα των συνεισηγητών. Καταρχήν υπάρχει μια ανάγκη για απλοποίηση και διευκρίνηση του κειμένου. Γι' αυτό θα πρέπει να αποφεύγουμε παρόμοιες διατυπώσεις κάπως ασαφείς και αόριστες. Ε, κατά προτεραιότητα επενδύσεις, δράσεις κλειδιά, κερίες δράσεις, Έχουμε κάποια προβλήματα λόγω της ασάφειας αυτών των όρων και άμα έχουμε προβλήματα εμείς φαντάζομαι ότι οι απλοί πολίτες ε, θα βρίσκουν ακόμη πιο δυσανάγνωστο το κείμενο όταν περιέχει τόσο προσδιορίστες έννοιες. Οι συμβάσεις εταιρική σχέσης δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ένα κατάλογο πόλεων για την επιδότηση του 5%. Συμφωνώ με τους συνεισηγητές εμείς να ορίζουμε μόνο τα κριτήρια, τις συνθήκες, αλλά να μην προβάλλουμε και ένα κατάλογο των πόλεων. Ένα άλλο θέμα είναι ο ρυθμός των μηχανισμών που υπάρχουν για την, Ευρω... για την περιφερειακή ανάπτυξη. Επενδύσεις, Τοπικέ καινοτομία κτλ. Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά του μηχανισμού, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα περιθώριο λιγμών για τα κράτη-μέλη, για να μπορούν να αποφασίσουν πότε, που και πώ θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα επιμέρους εργαλεία και μηχανισμούς. Ένα άλλο θέμα που αφορά επίσης την ελαστικότητα που απαιτείται για τα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαμε τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης, τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης, να τις χωρίζουμε, οπότε οι αλλαγές να μην χρειάζεται κάθε φορά να εξετάζονται από την Επιτροπή. Θα πρέπει να έχουμε ένα, τον πυρήνα της σύμβασης που θα, τη χάνει, θα είναι το αντικείμενο διαπραγμάτευση με την Επιτροπή, αλλά θα υπάρχει και ένα τμήμα που θα είναι πολύ πιο ελαστικό και θα μπορεί να ε, υπάγεται πολύ πιο εύκολα σε αλλαγές χωρίς να επαναλαμβάνουμε την επαχθή διαδικασία. Επίσης, ε, έχουμε πολλά σημαντικά επενδυτικά προγράμματα που απαιτούν χρονοβόρα διαδικασία. Υπάρχουν πολλές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, για παράδειγμα. Και πολλές φορές οι διοικητική διατυπώσεις είναι ιδιαίτερα επαχθής. Ε, στο μέλλον, λοιπόν, χρειάζεται να φροντίσουμε μια, για μια πλούστευση. Τελευταία μου ερώτηση αφορά τα 10 εκατομμύρια του μέσου της διευκόλυνσης ε, συνδέοντας την Ευρώπη, του Connecting Europe. Δεν συμφωνώ με την πρόταση αυτή, γιατί πιστεύω ότι έτσι θα περικοπούν κονδύλια από τη πολιτική συνοχή που είναι απολύτω απαραίτητα. Η Κωνσταντσα Κρέλ ξαναζήτησε το λόγο για ένα σχόλιο. Συγγνώμη, αλλά ξέχασα τελείως την τροπολογία για τον προπολογισμό. που είναι ίσως από τις πιο ενδιαφέρουσε τροπολογίε που έχουν υποβληθεί. Το είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Αυτό που έγινε είναι για όλα τα νούμερα της πρώτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάζουμε ένα χ και τα τροποποιούμε γιατί θέλουμε να διευκρινίσουμε όπως λέμε και στην αιτιολόγηση ότι μας δεσμεύει η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως αναφέρεται στην έκθεση Γκαρίγκα. Δηλαδή, Θέλουμε αύξηση του προπολογισμού Και αναφέρεται στην έκθεση Γκαρίγα ότι ακόμη και με αύξηση του επίπεδου πόρων για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό ταμείο χρειάζεται ένα 5% σχέση με το 2013 και παρόλα αυτά ένα μικρό τμήμα θα συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην αρχή της Ευρωπαϊκής Ελληνικής. Ως εκ τούτου θέλουμε τουλάχιστον να αύξη κατά 5% των πόρων για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα για την πολιτική συνοχή. Εκεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να διατηρηθεί τουλάχιστον ε, στα επίπεδα της περίοδου 2007-2013. Δηλαδή 366,2 ε, ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Χωρίς το CF. Αυτό το αναφέρουμε και στην αιτιολόγηση. Αν λοιπόν καταφέρουμε στις διαπραγματεύσεις ε, να γίνει δεκτό ο προπολογισμό που προτείνουμε, θα έχουμε ακόμη περισσότερα κονδύλια από ό,τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, πρότασή τη. Και στο πλαίσιο αυτό είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί η χρηματοδότηση και για τις ε, αξιόχως απόκεντρες περιοχές. ή να προβλέψουμε ένα δίκτυο ασφαλείας για τις ε, περιοχές μετάβασης. Ε, αλλά εκεί ίσως χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια, θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Προς το παρόν περιλαμβάνεται μόνο στη αιτιολογία. Είπαμε να μην κατατεθούν άλλες δημοσιονομικές τροπολογίες, άλλες τροπολογίες για τον προϋπολογισμό στην πρόταση. Γιατί θα, από τη στιγμή που δεν έχουμε απόφαση οριστική για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο θα απορριφθούν. Αυτά ως προς το υπέροχο άρθρο 84. Και θα αντιλαμβάνεστε γιατί έγιναν όλες αυτές οι προσπάθειες. Πάντως, επαναλαμβάνω, ευθυγραμμιζόμαστε με την ε, ομάδα διαπραγμάτευσης για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, Μπέγκε και λοιπούς. Και συμφωνούν με την κατεύθυνση αυτή. Ο κύριος Γκοτσμάνης. Ευχαριστώ. Μόλις ήρθα από την Επιτροπή Προπολογισμών όπου είμαι πλήρες μέλος. Τακτικό μέλο και ήθελα να πω ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, όχι μόνο για το επόμενο δημοσιονομικό, πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και για την ε, επόμενη χρονιά. Θα πρέπει για τη συνοχή να έχουμε διψήφιο ρυθμό ανάπτυξη και τέτοιε προβλέψει θα πρέπει να μα βρίσκουν επιφυλακτικού το Συμβούλιο συμφωνεί με προτάσεις της Επιτροπής. Αυτό θα ήταν λοιπόν ένα πρώτο βήμα να έχουμε μια τέτοια αύξηση για τον επόμενο προπολογισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις πληρωμές της συνοχής και όπως είπε και ο Επίτροπος Λεβαντόφσκι, μιλάμε για νόμιμες, θεμητές πληρωμές. Βέβαια, κάποιοι λένε δεν μας νοιάζουν αυτά. 200 δις τα έχουμε, δεν υπάρχει θέμα αν δεν γίνουν όλε οι Εγώ όμω νομίζω ότι μπορεί να γίνει πολύ σοβαρή κατάσταση ό,τι αφορά και την επόμενη περίοδο προγραμματισμού, το επόμενο πολιετέ πλαίσιο. Διαβάζω πολύ προσεκτικά τι ε, προτάσει που έκαναν οι εισηγητέ. Και λίγο πολύ μπορώ να συμφωνήσω με όσα έχουν ε, περιλάβει στον γραφό του. Όμω επιμένω στην πρότασή μου. Επιμένω και αναφέρομαι εδώ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ακόμη και στην περίπτωση που θα πάρουμε λιγότερα κονδύλια, αυτό δεν είναι λόγο να υπαναχωρήσουμε σε σχέση με τι αρχέ μα που έχουν καταγραφεί στον κανονισμό 1083 στο παράρτημα 2. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητε των επιμέρου περιοχών και χωρών και όχι να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, διακριτική μεταχείριση στην, ε, στα όρια που θα που θα τεθούν και τις διάφορες περιοχές. Για τις ε, περιοχές 3, που 3 ε, έχουμε ένα όριο από το 3,2 στο 3,7. Εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε διαλλακτικότητα και ευελιξία. Αυτό το προασπίστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν πρέπει να απομακρυνθούμε από τις αρχές μας, ακόμη και αν οι διαπραγματεύσεις είναι πολύ σκληρές. Νομίζω το τι θα ε, συζητηθεί στα πλαίσια του επόμενου προπολογισμού της επόμενης χρονιά θα καθορίσει και το επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστούμε. Για την ΚΟΑ, η κυρία Κονέλη. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να πω τα εξής. Στις νέες ε, προτάσεις, ε, στις νέες τροπολογίες βλέπω πολύ θετικό το ζήτημα των ε, εταιρικών σχέσεων, των συμβάσεων σχέσεων, σχέσης, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάσετε, η προσέγγιση, η ιδιαίτερη προσέγγιση στα άτομα με ειδικέ ε, ανάγκε, με αναπηρίε. Όλα αυτά πολύ καλά. Για τα, για τα χρηματοοικονομικά μέσα όμως. Υπάρχουν διάφορες τροπολογίες, 88 και 90 Φερρυπίν. Και εδώ θα ήθελα να παρακαλέσω τους δύο συνεισηγητές να μας εξηγήσουν τι ακριβώς εννοούν και τι αποσκοπούν με αυτό. Γιατί ναι, εγώ βλέπω ότι καλά είναι τα δημοσιονομικά μέσα, αλλά πού θα εφαρμοστούν κατά κύριο λόγο ή κατά προτίμηση. Η Επιτροπή πώς μπορεί να επηρεάσει την εξέλιξη και πώς μπορεί να εγγραφεί αυτό στο κείμενο της, ε, ε, του κανονισμού. Εάν έχουμε κατεξουσιοδότηση πράξης, τι υλοποίηση θα έχει αυτή η διάταξη, αυτή η πρόταση. Αυτό λοιπόν γιατί είναι ξεκάθαρο. Και δεύτερον, τα ποσοστιαία που δώσατε. Νομίζω ότι Τώρα με την εγκατάλειψη των ποσοστιαίων στοιχείων, Φερρυπίνη 94, άρθρο 94, η κατάσταση γίνεται αρκετά συναρπαστική θα έλεγα. Διότι μπορεί να υποκρύπτεται ο κίνδυνος, και εδώ αναφέρομαι σε προτάσεις με τη Γερμανία υπόψη και τη Φερρυπίνη η γερμανική κυβέρνηση νομίζω ότι είναι έτοιμη, διατεθειμένη προτάσεις ε, ή μάλλον κονδύλια που ενδεχομένως να ζητούσε στο ε, μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα προβλέψει σε μια ανάκρη για να τα έχει διαθέσιμα όποτε χρειαστεί. Εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι μπορούμε τόσο νωρί ή τόσο άμεσα να περάσουμε κατευθείαν στο 5%. Τακτικά τουλάχιστον θα θεωρούσα ότι ήταν εσφαλμένη προσέγγιση. Για το κοινό πλαίσιο αναφορά, εντάξει, δεν έχω αντίρρηση. Αλλά θα δούμε τι εφαρμογή θα δει, θα έχει. Γιατί πολλές φορές ε, εύκολο να λες κάτι που εδώ να το εφαρμόζεις. Και άλλη ερώτηση, υπάρχουν ενόψει και άλλες τροπολογίες ή πώς θα το χειριστούμε το θέμα, Εάν κάτι λείπει, τι θα κάνουμε. Ζητήματα περισσότερο γραφειοκρατικά, πιστοποίηση, αναγνώριση, συμμετοχή κτλ. Πώς θα αντιμετωπιστούν αυτά ή έχει κλείσει ο κύκλος των τροπολογιών και δεν υπάρχουν άλλες. Και ακόμη κάτι το οποίο το λέω κάπως αυθόρμητα και απροετοιμάστα, ότι αισθανόμαι μεγάλες ανησυχίες για τις ε, περιφέρειες που βρίσκονται σε μετάβαση, ιδιαίτερες ανησυχίες θα έλεγα, όχι απλώς ανησυχίες, και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πιστεύω το τι ακριβώς ζητούμε, το τι ακριβώς θέλουμε και να εμείνουμε σε αυτό, διότι στην ε, διάρκεια όλων αυτών των χρηματοοικονομικών διαπραγματεύσεων πολλές είναι οι ανησυχίες που αισθάνομαι, πολλά είναι τα αδύνατα σημεία που διακυγνώσκω, και ενδέχεται το πρόβλημα να ε, διαδοθεί περισσότερο. Αλλά δεν μπορώ να δώσω πιο συγκεκριμένους όρους, δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά, πιο απτά. Απλώς ρωτώ με αρκούν αυτά που λέει η Επιτροπή. Επιτρέψτε μου να αμφιβάλλω. Είναι ένας προβληματισμός δικός μου, εσωτερικός λίγο πολύ. Αλλά δεν αισθάνομαι ήσυχη με τις προτάσεις που έχω δει από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ την κυρία Ένστ. Δεν την έχω ξαναδεί τόσο πολύ να την απασχολεί κάτι και να θέλει να συμμετάσχει τόσο ενεργά. Με προσωπική παρέμβαση λοιπόν κύριε Πίπερ. Φαντάζομαι ότι και εσείς όπως συνήθως οι Γερμανοί θα είστε πολύ συναισθηματικός στην παρέμβασή σας. Ναι, δεν μπορώ αυτό να το πω σε σχέση με τη μεταβατική κυβέρνηση. Μπορώ να σας απαντήσω κυρία Έρνστ. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε και πάλι. Δυστυχώ τα σχόλια δεν ακούγεται. ακούγονται. Ε, Πάντω, φοβόμαι ότι ίσω να μην σα αρέσει η κατεύθυνση μπορεί να λάβει η εξέλιξη, διότι εμείς τροπολογίστε θα καταθέσουμε οπωσδήποτε. Αγαπητή Κωνσταντσε Κρέλ, μην ανησυχεί. δεν είμαι ο μόνο. δεν είμαι ο μόνο. Ο Γιάννου Ούλμπριχτ επίση χαίρεται ιδιαίτερη ικανοποίηση. Α, τώρα βλέπω ότι πρέπει να σοβαρευτούμε. Τρία-τέσσερα σημεία θα ήθελα να δω και τα λέω πολύ επιγραμματικά. Καταρχά. για τη δέσμευση των κονδυλίων. Θα ήθελα, δεδομένου ότι προέρχομαι και από πιο πλούσια, πιο ευμαρή περιφέρεια, να πω ότι δεν αντιλαμβάνομαι πώς είναι δυνατόν να πρέπει να χρηματοδοτήσουμε το 52% των κονδυλίων από το κοινωνικό ταμείο. Νομίζω ότι είναι ασφαλμένη αυτή η προσέγγιση. Χρειάζεται περισσότερη ευελιξία. Και χρειάζεται να κοιτάξουν πιο προσεκτικά αυτό που θέλουν οι ίδιες περιφέρειες. Όχι αυτό που έχει ορίσει για το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τα άλλα συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά τα οποία καταγράφουν στις προτάσεις τους οι συνεισηγητές που αποτελούν πιστεύω το 80 και θέσεις του Κοινοβουλίου. Αλλά θα ήθελα να συζητήσουμε πολύ πιο προσεκτικά το θέμα της μεταφοράς επιχειρήσεων ή παραγωγικών μονάδων είναι ένα θέμα που σας έχει απασχολήσει ιδιαίτερα και πιο, πολύ, πιο παλιά στι προηγούμενε αιτίε, Είναι ένα θέμα που προξενεί ε, πολύ μεγάλη δυσφορία και άρα θα πρέπει να καταθέσουμε τι σχετικέ τροπολογίε, πιστεύω. Για τον κύριο Κλάζακ θα ήθελα να πω ότι εάν αυτό το Connecting Europe ε, Facility, αυτά 10 δισεκατομμύρια δηλαδή, τα οποία ε, μπαίνουν στο Connecting Europe Facility, στο μέσο συνδέοντας την Ευρώπη δηλαδή, από τη συνοχή και τα επικρίνεται Εάν διατυπώνεται επικρίσεις εις βάρος αυτού του μέσου, νομίζω ότι κάνετε λάθος, γιατί νομίζω ότι θα έπρεπε να υποστηρίζουμε τα, τις περιφέρειες, τα κονδύλια αυτά, θα έπρεπε να υποστηρίζουμε το Connecting Europe και το Ταμείο Συνοχής. Ιδάλλως, ούτως ή άλλως θα χαθούν τα χρήματα, θα γυρίσουν πουθενά σε, σε άλλους κορβανάδες. Ας είμαστε ρεαλιστές. Το ότι δεν υπάρχουν αριθμητικά στοιχεία, εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου, κύριε Έρνστ νομίζω ότι είναι η πιο σωστή στρατηγικά και διαπραγματευτικά τακτική. Θα ήθελα να πω το εξή τώρα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά, όπως άλλωστε και σε πολλά άλλα μεγάλα ευρωπαϊκά κράτη. Ε, και τώρα με την ε, πρόταση αυτού του κανονισμού για περισσότερα διευθυντικά μέσα μπορούμε να αποστείλουμε εμεί από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σαφή μηνύματα. Εγώ λοιπόν υπογραμμίζω ήταν την ανάγκη για επενδύσει για την ανάπτυξη, για ε, υποστήριξη νέων επιχειρηματικών δράσεων, για ε, υποστήριξη υποδομών που θα έχουν ε, αντίκτυπο στην πραγματική, στην καθημερινή ζωή του πολίτη. Έτσι ώστε να βοηθήσουμε αυτές τις περιφέρειες. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω στο κείμενο είναι μάλλον business as usual, σαν να μην έχει γίνει τίποτα, ενώ έχουν αλλάξει τα πάντα, έχει αλλάξει η Ευρώπη, μετα, μεταλλάσσεται η Ευρώπη και δεν μπορώ να περιοριστώ μόνο στους, ε, ε, στην εικόνα που δίνουν τα κράτη Friends of Better Spending σε επίπεδο συμβουλίου. Θα πρέπει να δούμε και εμείς στο Κοινοβούλιο πώς θα τοποθετηθούμε και βεβαίως ήδη η πολιτική μου ομάδα σε ένα βαθμό έχει τοποθετηθεί. Ε, υποστηρίζουμε όμως πάντα και θέλω να το υπογραμμίσω πολύ καλύτερη υποστήριξη της ανάπτυξης. Επίσης, ε, στο θέμα του ε, μέσου για την ε, σύνδεση της Ευρώπης, δέοντας την Ευρώπη και το συσχετισμό με το Ταμείο Συνοχής. Ιδιαίτερα στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, εκεί που υπάρχουν τα μεγαλύτερα ελλείμματα, οι μικρότερες δυνατότητες επικοινωνίας, νομίζω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε ιδιαίτερα τις υποδομές και αυτό είναι κάτι το οποίο σε συνεργασία με την ομάδα μου ε, θα διατυπώσω τροπολογίες. Άλλωστε αποτελεί αυτό κεντρικό αίτημα και της δικής μου εκθέσεως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Μαρίτα Σάντσο Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πολύ γρήγορα να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές για αυτό το σχέδιο έκθεσης που πραγματικά αντικατοπτρίζει τις πολυάριθμες συζητήσει που είχαμε εδώ και μήνες. Πολύ γρήγορα να σταθώ σε δύο-τρία σημεία. Πρώτα απ' όλα η σημασία να μην διαγραφεί πλήρω το άρθρο 21 για την αιρεσιμότητα, τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Καλό θα ήταν να εμπνευστούμε από όσα είδαμε το πρωί και από τις προτάσεις της ΕΑΠΕΜ και αναλόγως να προγραμματίσουμε τις πιστώσεις. Χάρη στην επόμενη πολιτική περιφερειακή ανάπτυξη. θα πρέπει τα κονδύλια που θα εκταμιευθούν να ε, κατευθυνθούν σε επενδύσεις με ευρωπαϊκούς στόχους. Ως προς την αριθμότητα των δαπανών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ε, διευκρινίσει το καθεστώς ειδικών επιδοτήσεων για την επόμενη φάση της εδαφικής ε, Συνεργασία και ανάπτυξης προκειμένου να μην υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό. Επίσης, θα ήθελα να γνωρίζω τις συνολικέ δαπάνε για τα ταμεία, τα περιφερειακά ταμεία και το πώ θα κατανεμηθούν οι πιστώσεις της εδαφικής συνεργασίας αναπρόγραμμα, όχι ανακρατός μέλος, ώστε να μην υπάρχει ε, ε, ανισόρροπη εθνική κατανομή και θα πρέπει επίση να υπολογίσουμε σωστά και την επιστροφή των επενδύσεων και για την, και για, τροπολογία, για την τροπολογία που αναφέρει τι επενδύσει 122 μάλλον, που αναφέρει τι επενδύσει εκτό προγραμμάτων. Εδώ υπήρχε ένα όριο, ανώτατο όριο 10%. Κάτι προσθέθηκε όμως στην τροπολογία αυτή. Ένα ελάχιστο 1% στήριξης από το Ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης εκτός προγράμματος. They, they took from me. Ε, νομίζω αυτός ήταν ο κατάλογος των αγορετών. Ε, κυρία Γουκατσέφσκα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ θερμότατα και την Κωνσταντσα και τον Λάμπερτ γιατί σίγουρα η έκθεσή τους δεν είναι καθόλου απλή, το έργο τους δεν είναι καθόλου εύκολο και από τις παρατηρήσεις ε, διαπιστώνουμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, υπάρχει δυνατότητα για κανονισμό που να ικανοποιεί τους πάντες, που να καλύπτει όλες τις επιθυμίες ή που να διασκεδάζει όλες τις ανησυχίες. Πάντως συμφωνώ με τις περισσότερες τροπολογίες. Εγώ είμαι υπέρμαχος της μεγαλύτερης ελαστικότητας, της λιγότερης γραφειοκρατίας και ελπίζω ο κανονισμός να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Δεν συμφωνώ με τον Μάρκους Πίπερ που λέει ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να συμφωνήσουμε, ότι σώνει και καλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Αυτό το ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε, για μένα αυτή είναι η υποχρέωση είναι αδιανόητη. Θα οφείλαμε, θα μπορούσαμε, καλά, αλλά όχι ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να συμφωνήσουμε, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε. Προτιμώ να ευθύσουμε μια πιο ήπια διατύπωση, γιατί υπάρχουν πολλοί που έχουν αμφιβολίες και διαρωτώνται κατά πόσο αυτά τα 10 δισεκατομμύρια θα πρέπει να τα βγάλουμε από το Ταμείο συνοχή. Πάντως είμαι πεπισμένη ότι πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν, κατα... δεν θα καταφέρουν να εκταμιεύσουν τέτοια τα κονδύλια αυτά. Εγώ είμαι υπέρ ε, της ε, διαχείρισης ε, στη βάση και όχι εκ των κατανομή. Έχω πολλές αφιβολίες γιατί δεν υπάρχουν εθνικοί εθνικά πακέτα και για πολλές χώρες ε, θα είναι δύσκολο να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη, του Connecting Europe. Προτιμώ να γίνεται μια διαχείριση περισσότερο τοπική, περιφερειακή. Ένα άλλο θέμα που δεν έχει αναφερθεί. Εσείς ε, τι γνώμη έχετε, συμφωνείτε με τον Μάρκους Πίπερο ότι θα πρέπει χωρίς όρους ε, αυτό το κονδύλιο του τομείου Συνεχής να απομακρυνθεί ο κύριος Βίκτορ Μποστινάρου. Ευχαριστώ. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Θα αναφερθώ σε αυτό το, το CF χωρίς αριθμούς όμως. Πάντως είναι προφανές ότι η αρχή που πρότεινε ο κύριος Πίπερ αν σας αρέσει αλλιώς ξεχάστε το, δεν νομίζω ότι είναι λογική, ειδικά για το CF. Και τώρα, αν θα πρέπει να πούμε ή θα δεχτείτε τη μεταφορά ή θα, χάσετε δισεκατομμύρια ευρώ, αυτή η προσέγγιση είναι πολύ άδικη γιατί θα τροποποιήσει ριζικά το κάπινγκ, το ανώτατο όριο, γιατί Κάτι τέτοιο θα πλήξει κέρια όλο το θέμα της κατανομής των κονδυλίων της συνοχής. Γιατί ποιο κράτος μέλος από το Συμβούλιο θα δεχτεί ε, νέα συζήτηση για το κάπινγκ, για τον προσδιορισμό των ανωτάτων ορίων. Αυτή η δυνατότητα μεταφοράς των 10 δισεκατομμυρίων θα ε, μειώσει δραματικά τα εθνικά πακέτα τους τα, τους εθνικού, τα εθνικά ποσά. Εγώ είμαι υπέρ του ΣΥΕΦ, εγώ είμαι υπέρ της εφαρμογής τέτοιων σχεδίων που είναι υποφελή για την Ευρώπη, που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των κρατών μελών και τις ανησυχίες των Ευρωβουλευτών και προσπαθούν να βρουν την απαραίτητη ελαστικότητα και την καλύτερη στρατηγική διεξόδου. Το, το take it or leave it νομίζω ότι δείχνει μια διαλαξία και θα επιτείνει την απογοήτευση, τη δυσφορία και ουσιαστικά θα ναυαγίσει όλο το σχέδιο του ΣΥΕΦ. Αν θέλουμε κάτι τέτοιο, εντάξει, αυτή η πιο διάλεκτη στάση, αν σας αρέσει, αλλιώς το ξεχνάμε, τότε μπορούμε να την υιοθετήσουμε. Πάντως δεν νομίζω ότι είναι αυτή η σωστή μέθοδος. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι εύλογε κατά τη γνώμη μου ανησυχίε πολλών χωρών. Δεν νομίζω ότι οι ανησυχίε αυτέ είναι ανέντιμες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρυσόγελος. Ήθελα, απλώ απλώς να τονίσω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε η κρίση έχει αλλάξει τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτόμαστε και πώς θα είναι το μέλλον τα επόμενα χρόνια. Άρα τα εργαλεία που συζητάμε δεν είναι κάτι το οποίο ανταποκρίνεται σε συνθήκες που ήταν μερικά χρόνια πριν, αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε πώ θα είναι οι συνθήκες μερικά χρόνια μετά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσουμε. Δηλαδή, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, εάν τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε είναι μια προηγούμενη περίοδου που δεν υπήρχε κρίση, σήμερα αυτά μπορούν να έχουν ανατραπεί πλήρω. Και αυτό το λέω σαν γενική αρχή για να το έχουμε υπόψη. Αν σήμερα μιλάμε ότι η απασχόληση είναι ένα πολύ κέριο πρόβλημα και βλέπετε τι γίνεται με την οργή που αναπτύσσεται σε διάφορες χώρες. Πρέπει στις πολιτικές των ταμείων είτε άμεσα είτε έμεσα να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη το θέμα της απασχόλησης, δημιουργία πραγματικά θέσεων απασχόλησης. Και αυτό πρέπει να προσδιορίσει λίγο και τις προτεραιότητές μας. Εάν δεν δώσουμε ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να απασχοληθούν, όλα τα άλλα που συζητάμε δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα και θα δημιουργείται μια αυξανόμενη ευρωσκεπτικότητα. Βλέπετε στην Ελλάδα ότι μπήκανε πολύ ακραίε δυνάμει στο Κοινοβούλιο που πριν μερικά χρόνια ήταν αδιανόητο για την Ελλάδα. Και όμω τώρα αυτή η οργή, γιατί οι πολίτε δεν βλέπουν αποτέλεσμα στη ζωή του. Και νομίζω το είπε καλά κάποιο προηγούμενο ε, εισηγητή, ότι πρέπει να φαίνεται και αποτέλεσμα στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Να μην μιλάμε μόνο με υποδομέ, μόνο με μεγάλα έργα, μόνο αφηρημένα νούμερα. Και το έχουμε συστήσει και παρόλο είμαι νέο εδώ στο Κοινοβούλιο, το ακούω συνέχεια να επαναλαμβάνεται και, το, την έννοια τη αποτελεσματικότητα. Αλλά η αποτελεσματικότητα δεν είναι μόνο ένα θέμα που έχει να κάνει με χιλιόμετρα ή απορρόφηση κονδυλίων, αλλά έχει να κάνει και πραγματικά να πετυχαίνουμε του ουσιαστικού στόχου. Τι σημαίνει περιφερειακή ανάπτυξη, τι σημαίνει κοινωνική συνοχή, τι σημαίνει περιβάλλον και πώς πράγματι επιτυγχάνονται και πώς μετριώνται αυτές οι επιτυχίες όταν διαθέτουμε ευρωπαϊκούς πόρους, πώς αυτά ε, μετριώνται και πραγματικά η κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι δεν σπαταλιώνται για να γίνει ένα έργο που μετά δεν χρησιμοποιείται. Και για να κλείσω, αναφέρω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα χρηματοδοτήθηκε η σιδηροδρομική υποδομή σε ένα ορισμένο βαθμό. Μέσα στι πολιτικέ που προωθήθηκαν και από την Κομισιόν ήταν πολλέ αυτέ οι γραμμέ να κλείσουν. Μα γιατί δώσαμε όμω τα χρήματα, οι Ευρωπαίοι πολίτε, γιατί δώσαν τα χρήματα αναφέρονταν ότι οι γραμμέ είναι βιώσιμε και αντί να κάνουμε βιώσιμε υποδομέ, περικόψαμε και δημοσιονομικού λόγου. Το ίδιο ισχύει και πολλά άλλα έργα. Άρα λοιπόν πρέπει να τα λάβουμε αυτά υπόψη πολύ σοβαρά και να, στον μελλοντικό σχεδιασμό να διορθώσουμε τέτοια θέματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Θα είμαι λακωνικός για ορισμένα θέματα του κανονισμού που χρήζουν στήριξη και πολύ σωστά τα αναφέρουν οι συνεισηγητές στην πολύ αξιόλογη έκθεσή τους και τις ε, σημαντικές τροπολογίες για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Άλλωστε αυτό είχαμε ζητήσει και εμείς και χαίρομαι που συμπεριλήφθηκε αυτό το θέμα. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την, ε, το υποχρεωτικό αποθεματικό επίδοσης στην Πολωνία είχαμε πολύ θετική εμπειρία με αυτό για πολλές περιφέρειες. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να ταχθούμε να αναφαδόν υπέρ αυτής της πρότασης. Τώρα, μία λέξη κλειδί για τον κανονισμό είναι η ελαστικότητα ελαστικότητα για το πώς θα διαθέτουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές τα κονδύλια ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις ιδιαιτερότητές τους. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι κλειδί αυτή η ελαστικότητα στον κανονισμό. Υπάρχουν όμως ε, μερικά θέματα που με προβληματίζουν κάπως ε, και μου δημιουργούν ανησυχίες. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε από τον κανονισμό να αφαιρέσουν οποιασδήποτε αλλαγέ του συστήματο διόρθωση. Ε, νέτο των καθαρών διορθώσεων. Νομίζω ότι αυτό το θέμα μπορεί κάλλιστα να διαγραφεί από τον κανονισμό, γιατί αποδυναμώνει την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδύλιων από τι ε, νέε κυρίως χώρε μέλη. Και νομίζω ότι δεν είναι σωστή αυτή η πρόταση και σε καμία περίπτωση δεν θα διευκολύνει την εκταμείευση των κοινοτικών κονδυλίων από τις χώρες δικαιούχους. Σε ό,τι αφορά ε, την πρόταση του κυρίου Πίπερ. Κατά τη γνώμη μου είναι τελείω ε, ανεδαφική αυτή η πρόταση. Να βγάλουμε τα ε, κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής και να τα μεταφέρουμε στο μέσο διευκολύνοντας την Ευρώπη, ε, την Ευρώπη, συγγνώμη, διευκόλυνση Ευρώπη, δεν νομίζω ότι ε, είναι σκόπιμο, γιατί ούτως ή άλλως αυτά τα κονδύλια θα αποφασίζονται στην Ευρώπη, δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα προσαρμογής ε, στις τοπικές ανάγκες, στις εθνικές ανάγκες των χωρών δικαιούχων. Είναι τελείως ανεδαφική, άστοχη αυτή η πρόταση της μεταφοράς και δεν συμφωνώ σε καμία περίπτωση ότι οπωσδήποτε, σαν και, καλά, και καλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε. Αντίθετα, θα πρέπει να στείλουμε μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και παραλαμβάνω εδώ αυτό που είχα πει και στην προηγούμενη μας συνεδρίαση όταν συζητήσαμε αυτό το θέμα με τον εισηγητή. Ότι σε κα... <laughs> Το αντίθετο, δεν πρέπει να συμφωνήσουμε. Η μεταφορά κονδυλίων από το Ταμείο Συνοχής στο μέσο συνδέοντος στην Ευρώπη είναι, ε, η πρόταση αυτή είναι ανόητη και τελείως αναδαφική. Νομίζω ότι τέτοιου είδου προτάσεις ε, σε καμία περίπτωση δεν θα ωφελήσουν, ε, γιατί είναι τελείως άστοχο, επαναλαμβάνω, μεταφερθούν κονδύλια από το Ταμείο Συνοχής στο συνδέοντα στην Ευρώπη, στο Connecting Europe. Κύριε Κλέβα, ευχαριστώ και εγώ να συγχαρώ τους συνεισηγητέ για το σχέδιο έκθεση, επειδή ετοιμάζω την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειών ε, για το θέμα της χρήσης αυτών των μηχανισμών ε, στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, με ενδιαφέρει ακριβώ ε, το σημείο των χρηματοδοτικών μέσων που περιλαμβάνει και καλύπτει η έκθεση αυτή. Είναι πολύ σημαντική η εξάρτητη αποτίμηση εδώ για να αντιμετωπίζουμε τις περιπτώσεις των αποτυχιών στην αγορά. Για την κατάσταση των επενδύσεων θα συμφωνήσω με όσα είπε η Κωνσταντσα Κρέλ ότι πρέπει να υπάρχουν σαφείς κανόνες, ιδίω στις πρωτογενείς πράξεις, σε αυτό το επίπεδο και όχι τόσο στις είναι αυτό είναι δική μου έκκληση. Επίσης καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβλέψει απαιτήσει για το ρόλο και την εφαρμογή της εξάντια αποτίμησης στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού, ιδίω μετά από όσα άκουσα και σήμερα το πρωί από τους εκπροσώπους των πόλεων, των αστικών κέντρων και του βασικού φορεί που ακριβώ θα χρησιμοποιήσουν τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα για δημόσιε διαδικασίε. Θα πρέπει τα χρηματοδοτικά αυτά μέσα να είναι ελκυστικά προ το κοινό, ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν. Νομίζω ο ρόλο του γενικού κανονισμού είναι να περιλάβει τουλάχιστον κάποιου γενικού αλλά απόλυτα σαφεί κανόνες. very... Θα πρέπει να είμαστε πολύ σύντομοι, γιατί όλο και μεγαλώνει ο κατάλογο των αγορητών. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και δεν ήθελα να ευχαριστήσω του ε, ομιλητές για τα όσα είπαν. Θα ήθελα να αναφερθώ όμως σε κάποιες πτυχές που μου φαίνονται πολύ σημαντικές. Τρία σημεία που έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Καταρχάς χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη ευελιξία κατά την επεξεργασία αυτών των ζητημάτων, σαφής ε, προτεραιότητε, αλλά από τη βάση προ τα άνω, από τις περιφέρειες δηλαδή προ τα άνω, όπως είπε και ο κύριος Μπίπολς, χρειάζεται μια συζήτηση για την δέσμευση των μέσων των κονδύλων, δηλαδή στο, ε, Ευρωπαϊκό, στο EFSF, ε, που δεν αποβαίνει πάντα σε όφελος των περιφερειών και θα ήθελα ιδιαίτερα για τη δική μου την ε, περιφέρεια στην Ανατολική Γερμανία να ζητήσω περισσότερη δυνατότητα προγραμματισμού, έγκαιρου προγραμματισμού και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Θα πρέπει να διευρυνθεί δηλαδή το δίκτυο ασφαλείας, το οποίο θα πρέπει να επεκταθεί και στις περιοχές που έχουν περάσει στο phasing out. Έχουμε περίπου 12 περιφέρειες, στο Νόμενο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, οι οποίες είναι στη φάση του phasing out και χρειάζεται προγραμματισμός. χρειάζεται να μπορούν να προγραμματίσουν τι είδου κονδύλια θα έχουν θέση του στο μέλλον. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστώ τους δύο εισηγητές. Ε, σημαντικά έχουν βελτιώσει την ε, αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την έχουν απλουστεύσει, και ίσως θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη, περισσότερη ε, βελτίωση. Θα πρέπει να προάγουμε την πολιτική συνοχή και τη διαφορετική πολιτική, όχι να την παρεμποδίζουμε με τις πολιτικές που εισάγονται. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε με εκπροσώπου των περιφερειών και των αστικών κέντρων που επίση ζήτησαν περισσότερη ευελιξία στα προγράμματά μας και άρα βλέπουμε ότι χρειάζεται να γίνουν αρκετά πράγματα με στόχο βέβαια τη στρατηγική 2020 αλλά και για την ανάπτυξη που πρέπει να, πρέπει να είναι ένα στόχος απτό ένα στόχο τον οποίο θα υλοποιήσουμε με τα μέσα των διαφορετικών ταμείων. Περίπτωση κατά την οποία, δεδομένου ότι οι περιφέρειε είναι αυτέ που γνωρίζουν καλύτερα τι χρειάζεται και πού χρειάζεται, πρέπει αυτέ να ε, είναι εκείνε που θα υλοποιήσουν τα μέτρα. Και βέβαια χρειάζονται και έργα υποδομών, με προτεραιότητε φυσικά που θα προσδιοριστούν. Έχω πει κάποιες ιδέες ώστε να προσθέσουμε και άλλες και σε, στο σημείο αυτό θα έπρεπε να προσδιορίσουμε μέτρα όπως το Connecting Europe που είναι συγκεκριμένο μέτρο επιγραμματικό ε, πρόγραμμα και άλλα αντίστοιχα με τις υποδομές ε, που μπορούμε να υποστηρίξουμε με παράλληλο στόχο και την ανάπτυξη απασχόλησης. Αγαπητέ Λάμπερτ, αγαπητή Κωνσταντζή, είναι πολύ καλή πρόταση. Σα ευχαριστώ πολύ και πιστεύω ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για μια πολύ καλή συζήτηση. Ο κύριος Ολεϊνίτσακ. Βόιτσεκ Μίχαου Ολεϊνίτσακ και όχι Βόιτσεκ Μάρεκ Ολεϊνίτσακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θεωρώ ότι ο κανονισμός αυτός ε, ε, και μάλλον η συγκεκριμένη έκθεση είναι ένα πολύ καλό σημείο αφετηρίας στα πλαίσια της ε, προετοιμασίας ε, και της διαμόρφωσης της πολιτικής συνοχής στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Χάρη στην έκθεση αυτή και στη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γίνει πιο ευανάγνωστη η πολιτική συνοχής πιο αποτελεσματική για όλους ε, τους δικαιούχους, για τη τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, για τους επιχειρηματίες, θα δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης. Όλα αυτά είναι τα ζητούμενα, οι επιθυμίες και οι στόχοι μας και περιλαμβάνονται στην έκθεση. Βέβαια, είναι πολύ πιο εύκολα αυτά τα θέματα για τη συνοχή από ό,τι για τη γεωρική πολιτική. Εκεί ε, αλλάζουν άρδινα ε, τα πράγματα. Έχουμε μια ρηξικέλευτη μεταρρύθμιση, οπότε η συζήτηση για την μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής είναι πολύ πιο περίπλοκη. Ενώ η αντίστοιχη συζήτηση για την πολιτική συνοχή είναι πολύ πιο εύκολη και υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση μεταξύ μα. Ελάχιστε είναι οι διαφορέ. Ε, μεταξύ μα σε σχέση με τι τεράστιε διαφορέ και διαστάσει απόψεων που υπάρχουν για τη μεταρρύθμιση τη κοινή αγροτική πολιτική. Ο διαξυφισμός με τον Μάρκο Πίπερ ε, είναι ασήμαντο σε σχέση με τι τεράστιε διαφορέ που υπάρχουν για τη γεωργική πολιτική. Το βέβαια το πιο επίμαχο θέμα εδώ είναι το θέμα του προπολογισμού και το μέσο Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη, είναι ένα πολύ καλό μέσο το CF είναι πολύ καλό και δεν ξέρω γιατί προκαλεί τέτοιου φόβου. Και μάλιστα και οι νέε χώρε μέλη θα μπορέσουν να υποφεληθούν από το Connecting Europe. Αυτό θα ήθελα να πω προ τον κύριο Πορέμπα και άλλου που έχουν δισταγμού. Τέτοιου είδου ε, μέσα όπω το Connecting Europe μα είναι χρήσιμα και στι νέε χώρε. Για παράδειγμα στι υποδομέ για του αγωγού φυσικού αερίου, για του ε, πετρελαγωγού, για τη δημιουργία, για την ε, κατασκευή εργοστασίων θερμοελεκτρικών και ούτω καθεξής τέτοιου είδους υποδομές μπορούν χάρη στο Connecting Europe να ολοκληρωθούν. Παρακαλώ, αν διαβάσετε προσεκτικά το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα δείτε ότι υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις που δίνουν ευκαιρίες και συμμετοχή στην διαδικασία λήψη αποφάσεων και στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, αλλά και στο μέλλον δίνονται τέτοιες εξουσίες ε, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για συμμετοχή στις διαβουλεύσεις. Οπότε για μένα δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το μέσο Connecting Europe. Φυσικά, αν είχαμε πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό ε, στην ε, πολιτική συνοχής, δεν θα χρειαζόταν να βγάλουμε κονδύλια από την πολιτική συνοχή για να τα πάμε στο μέσο Connecting Europe. Μακάρι να είχαμε περισσότερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει. Και εγώ είμαι κατά τη μεταφορά ε, του κονδύλιου αυτού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το μέσο Connecting Europe είναι κακό, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλό αυτό το μέσο. Ωραία. Τώρα θα ακούσουμε του δύο συνεισηγητέ. Ο Λάμπερτ. Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Εκτό και αν θέλει βέβαια εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει το λόγο. Δεν ξέρω αν οι συγητέ προτιμούν να ακούσουμε πρώτα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πίτερ, έχει σχόλια. Μερικά σχόλια για τις πρόσθετες τροπολογίες, όχι τις αρχικές. Υπάρχουν πολλά στοιχεία εδώ που θα μπορέσει να στηρίξει η Επιτροπή, όπως την εδαφική συνεργασία, την στήριξη των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες την αποτίμηση εξπόστ, τον ορίζοντα 2020. απλώς ένα θέμα για τα χρηματοδοτικά μέσα ήθελα να θέσω. Προτάθηκε να έχουμε περισσότερες λεπτομερείς τάξει, για το τι διευκρινήσει, τι στοιχεία θα περιέχουν κατά εξουσιοδότηση πράξη. Αυτό είμαστε ανοιχτοί. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι σε αυτή την εντολή εκχώρηση, σε αυτή τη ε, διαδικασία υπάρχουν όλε οι απαραίτητε λεπτομέρειε. Όσο για το ζήτημα τη εξάντε αποτίμηση. Κάποια στοιχεία θα μπορούσαν να τα περιλαμβάνει ο Γενικό Κανονισμό, όμω θα μπορούσαν για τι τεχνικέ λεπτομέρειε να καλύπτουν το θέμα οι κατεξουσιοδότηση πράξη σημειώνουμε το ερώτημα για το CSF και θα το σκεφτούμε. Απλώς δύο τελικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα για το 84-2, τα κριτήρια ρεσιμότητας και την εισαγωγή αναφορών σε δημοκρατικούς παράγοντες. Εδώ το θέμα είναι τεχνικού χαρακτήρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχούσε για το κατά πόσον τα στοιχεία που περιλαμβάνονται εδώ βασίζονται σε εναρμονισμένα δεδομένα για όλα τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν και δημογραφικές εξελίξεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οπότε γίνεται κάπως υποκειμενική όλη η προσπάθεια αξιολόγησης. Μια τελική παρατήρηση για το αποθεματικό επιδόσεων. Αυτό αναφέρθηκε και την περασμένη φορά. οι εισηγητέ διέγραψαν αυτό το απόθεμα επιδόσεων, αλλά και το άρθρο 20,4. Θα ήθελα να το σκεφτούν προσεκτικά. Το 20,4 Είναι η διατάξη που δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα να διορθώσει κάτι σε κάποιο πρόγραμμα, εφόσον έχει υπάρξει αποτυχία μερική ή πλήρης. Αυτό το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Όχι μόνο γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποχρεωθεί πολλάκι να το χρησιμοποιήσει, αλλά γιατί θα μπορεί να αποστείλει και ένα γερό μήνυμα όταν οι επιδόσει υπολείπονται των προσδοκιών. Θα ήθελα λοιπόν οι συγκεκριτές να το σκεφτούν. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ σύντομα τώρα οι συγκεκριτές. Κύριε Φανίστερβη. Ευχαριστώ πολύ για την ποικιλία των σχολείων. Τα έχουμε ακούσει κάποια αρκετές φορές όμως εδώ ακούμε και κάποιες νέες απόψεις. Είναι σημαντικό αυτό για να την πρόοδος. Όπως είπε η κυρία Ένστ, για τα χρηματοδοτικά μέσα, είναι σαφές χρησιμοποίησαμε κάποιες βασικές αρχές ώστε να υπάρχει σαφήνεια. Λόγω χάρη, αν να διαγραφεί το αποθεματικό επιδόσεων, αυτό σημαίνει ότι εφ' εξής, δεν μπορεί να χρησιμοποιείται πια το ποσοστό το 5% εφόσον διαγραφεί αυτό το τμήμα του κειμένου. Δεν θα χαθούν όμως αυτά τα κονδύλια. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία που θα μπορούσαν να αποσαφενιστούν περαιτέρω. Ρωτήσατε ποια είναι η κατάσταση της διαδικασίας αυτή τη στιγμή. Ήδη οι τροπολογίες έχουν περάσει για μετάφραση. Κάποιες πρόσθετε σήμερα ε, θα αποσταλούν ακριβώς για μετάφραση. Μόλις είναι έτοιμες θα τις έχετε στα γραφεία σας και θα μπορείτε και εσείς να κάνετε τα δικά σας σχόλια. Η Κωνσταντσε με ενημερώνει ότι για το CSF δεν υπάρχει διαδικασία από δική μας πλευράς. Τώρα για την ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την περασμένη φορά είπαν ότι για το CSF, το Ελληνικό Ταμείο, μπορούσε να σκεφτούν θα σκέφτονται μάλλον τι θα γίνει το μεταξύ. Τώρα θα σκεφτούν κι άλλο. Πολύ περισυλλογή έχει πέσει. Χρειαζόμαστε και κάποια πρόοδο. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιε καθυστερήσεις και παιχνίδια τακτική. Στην επαφή μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω πρέπει να καταστεί σαφές Χρειαζόμαστε έναν πυρογνώμονα να κοιτάξει το κείμενο να καλύψουμε τα όσα λένε ότι θα υπάρχει νομική πρόβλεψη εδώ με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει φρεθεί ώστε να μην χρειάζεται μεταδιαρκής αναθεώρηση, τεχνική αναθεώρηση. Άκουσα βεβαίως τη δική σας την ε, σκοπιά. Θέλετε να σκεφτείτε να συλλογιστείτε και μετά να προτείνετε. Ε, ναι, πολύ σύντομα και για τα το γιατί για τα οικονομικά μέσα, πρέπει οπωσδήποτε να προσδιορίσουμε κάποιου βασικού κανονισμού στον κανονισμό. Φυσικά δεν μπορούμε να προβλέψουμε κάθε διάταξη σε κάθε λεπτομέρεια και κάθε κατεξουσιοδότηση πράξη, αλλά κάποιε προποθέσει ή μη τι άλλο στο γενικό κανονισμό μπορούμε να τι ενσωματώσουμε. Και αυτό νομίζω αποσκοπούν και οι τροπολογίε που έχουμε καταρχά καταθέσει. Κάποιε επιπλέον θα υπάρξουν ασφαλώ και ο Λάμπερτ και εγώ οπωσδήποτε έω τι 29 Μαΐου θα ε, ασχοληθούμε με την προετοιμασία επιπλέον τροπολογιών, τις οποίες θα καταθέσουμε στην τακτική διαδικασία, όπως και οι λοιποί συνάδελφοι φαντάζομαι. Για τον... Ε, προπολογισμό και τις σχετικές τροπολογίες. Εμείς περιοριζόμαστε μόνο στα όσα έχει αποφασίσει η διάσκεψη των Προέδρων. Ευελιξία δεν έχουμε στο πεδίο αυτό, πολύ λίγοι και στην αιτιολόγηση προσπαθούμε να εξηγήσουμε ποια είναι η βάση πάνω στην οποία δρούμε και γιατί προβαίνουμε σε αυτή την επιλογή. Νομίζω ότι είναι πολύ εύστοχη και σωστή. Στο ερώτημα για την ευελιξία για τις περιφέρειες, δεν θέλω να πω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο έχουμε αναλάβει να εξετάσουμε σε προσεχή γύρω και με τις τροπολογίες μας. Είναι σαφές Ε, τέθη ζήτημα αν υπάρχει ανάγκη για περισσότερες προτεραιότητες και αν ε, μπορούσαμε να διατυπώσουμε και άλλες προτεραιότητες. Νομίζω ότι νομοτεχνικά θα ήταν πρόβλημα αυτό προς την ορθή διατύπωση δηλαδή του γενικού κανονισμού. Θα έπρεπε ενδεχομένω σε ειδικού κανονισμού, σε επιμέρους κανονισμούς να ενσωματωθούν αυτές οι προτάσεις και ο Γιάννης Φαλός ε, θα καταθέσει ως αρμόδιος ηγητής τις προτάσεις του στο θέμα αυτό για την μετακίνηση, μετατόπιση επιχειρήσεων τόπων παραγωγής ήδη προβλέπεται στον, σε άλλο κανονισμό, αλλά εάν νομίζετε ότι είναι πολύ σημαντικό, πολύ ευχαρίστω να το ενσωματώσουμε, είναι κάτι το οποίο ούτως ή έχει πάντοτε με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθήσει και κρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλάμε ήδη για ένα δεύτερο γύρο τροπολογιών, ωστόσο νομίζω ότι οι περισσότεροι από τους συναδέλφους αναφέρθηκαν ήδη στο μέσον συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe Facility. Και θα ήθελα να διατυπώσω την εξή παρατήρηση, ότι αντιλαμβάνομαι βεβαίω ότι θεωρούμε ότι με δεδομένη την ε, τωρινή κατάσταση είναι απαραίτητο να υπάρχουν αυτά τα μέσα για τα, κάθε κράτο. Αλλά σε μια παρατήρηση που έκαναν ε, κάποιοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι. Το να πιστεύουμε ότι μπορεί να ε, ο βότσε και να ότι μπορεί να χρησιμεύσει για την ανάπτυξη υποδομών, μεταφορών και λοιπόν υποδομών. Μην να σα υπενθυμίσω ότι εμείς πάντοτε αυτό υποστηρίζαμε ότι και υπογραμμίζαμε ότι σπάνια τα κράτη-μέλη δείχνουν ενδιαφέρον για υπερσυνοριακές υποδομές, για έργα υπερσυνοριακά. Απλώς κοιτούσαν έναν εύκολο τρόπο, ένα γρήγορο τρόπο να συνδεθεί μια πρωτεύουσα με την άλλη ενδεχομένω, από την μια περιφέρεια στην άλλη και αυτό ήταν όλο. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εξασφαλίσουμε συμμετοχή των κρατών μελών, ουσιαστική συμμετοχή, ώστε να μην επιβάλλεται άνωθεν η επιλογή αυτή. Νομίζω ότι το να, το να ανατρέψουμε την ιδέα αυτή θα ήταν πολύ εσφαλμένο. Θα ήταν σαν να και είχαμε τα, τα χλωρά με τα ξερά μαζί. Το strategic frame, το ε, στρατηγικό πλαίσιο, ναι, θα ήθελα να πω ότι έχουμε το άρθρο 20 παράρθρος 4 που θα πρέπει να επανεξετάσουμε. Μέχρι στιγμής αυτά μπορώ να σας πω μόνο. Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία, μια και έχουμε και την Προεδρία παρούσα σήμερα, να επισημάνω πολύ ξεκάθαρα ότι βεβαίως μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός, βεβαίως πολιτική συνοχής είναι δύο έννοιες συναφείς, αλληλοσυνδεόμενες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η διαπραγμάτευση του δημοσιονομικού πλησίου μπορεί να συνδεθεί με το μέσο το οποίο διαπραγματευόμαστε για την πολιτική συνοχή που υπάγεται στην διαδικασία της συναπόφασης. Βρισκόμαστε σε, μια αυστηρή, σε ένα αυστηρό διαχωρισμό των νομοθετημάτων. Δεν μπορεί να λέει το, το Συμβούλιο αυτό είναι το πακέτο, πάρτο ή έχεις χάσει τα πάντα. Όχι, διαφοροποιούνται, δεν περνάει αυτό που ζητάτε και δεν ήταν αυτό το νόημα της συνθήκης της Λισαβόνας και της σχετικής ε, καινοτομία που εισήγαγε με έγκριση από τα 27 κράτη-μέλη. Πρέπει να επισημάνω με την ε, πολιτική τη ε, διαδικασία συναπόφαση. Γι' αυτό λοιπόν μην προσπαθείτε να τα αναμίξετε όλοι. Πολιτική συνοχή συνεχίζει με τη διαδικασία της συναπόφασης και θα το υπενθυμίζουμε στο Συμβούλιο στις διαπραγματεύσεις μας, όπου ελπίζουμε ότι θα τύχουμε συνεργατικής αντιμετώπισης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Δυο λεπτά ακόμη θα σας ζητήσω υπομονή για να κλείσει όλη η συζήτηση. Κάποιος που μπορεί να κοιτάζει τα πράγματα από ψηλά και από απόσταση, σαν πουλί μπορεί να βλέπει πράγματα που δεν τα βλέπετε με τη μια. Όπω α πούμε την έμφαση που θέλουμε να δώσουμε από τη μια για τι τηλεπικοινωνίε και τι μεταφορέ και την συνεργασία και από την άλλη για την προστεθέμενη αξία τη μετατόπιση από τα 10 δισεκατομμύρια των εθνικών κονδυλίων προ το κεντρικό, προ την κεντρική διαχείριση. Εδώ πρέπει να δούμε κατά πόσον τα κονδύλια αυτά θα πλήξουν την ε, προστασία των εθνικών ιδιωτήτων. Θα πρέπει λοιπόν τα στοιχεία αυτά να τα δούμε παράλληλα. Εάν θέλουμε να έχουμε μια εμπεριστατωμένη άποψη ω Επιτροπή Ρέτζι τα θέματα αυτά. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για τη μετάφραση. Την ε, εβδομάδα αυτή θα έχουμε τι προηγούμενε τροπολογίε που έχετε ήδη αποστείλει και οι τωρινέ τροπολογίε αυτού του σχεδίου έκθεση θα είναι διαθέσιμε σε όλε τι γλώσσε το αργότερο 21 Μαΐου στο Στρασβούργο. Στις 21 Μαΐου λοιπόν. Νωρίτερα από την λήξη της προθεσμίας. Σε όλες τις γλώσσες. Δεύτερο σημείο για το CSF. Καταλαβαίνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το σκέφτεται. Αλλά χρήσιμο θα ήταν, και το παραλαμβάνω, γιατί θα αποφασίσει η Επιτροπή μα, να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να συντονιζόμαστε εδώ στο δυνατόν συντομότερα. Θέλουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση την καλύτερη δυνατή επιλογή. Ένα έγγραφο εργασία. Δύο, κάτι που να εντοπίζετε τι καλύτερε επιλογέ που θα πρέπει να συζητήσουμε. Και τα τρίτον, να πω ότι θεωρήσουμε προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών ω τι 31 Μαου 6 το απόγευμα από σήμερα. Καμία καθυστέρηση δεν θα συγχωρεθεί. 6 το απόγευμα 31 Μαΐου. Για μια προσωπική συμβουλή. Μέχρι το τέλος να παρακολουθείτε τις τροπολογίες που υποβάλλετε, διότι κάποιες φορές το σύστημα πληροφορικής μπλοκάρει και κάποια πράγματα χάνονται. Μην τα αφήσετε λοιπόν να ξεφύγουν από την προσοχή σας επίσης. Προθεσμία υποβολής τροπολογιών και για την έκθεση του κυρίου Μποστινάρου και για την έκθεση του κ. Τέλερ, που δεν θα συζητηθούν σήμερα. Και τελευταίο στοιχείο να σας θυμίσω ότι όλες οι τροπολογίες, με συγχωρείτε που είμαι τόσο αυταρχική ως πρόεδρος σήμερα, αλλά να σας θυμίσω ότι όλες οι τροπολογίες πρέπει να υποβληθούν ως προς την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι την έκθεση της Κωνσταντζα και του Λάμπερτ. Στην πρόταση τη Επιτροπή θέλουμε να προτείνουμε αλλαγέ. Να, προτείνουμε, να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο τη ημερήσια διάταξη, στο Γιάνν Ολμπριχτ. Γιάνν, νομίζω ότι σου δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω αγγλικά γιατί το κείμενο το έχω στα αγγλικά. Οπότε θα είναι πολύ πιο εύκολο και για μένα να σα εξηγήσω τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά την ε, τελευταία σα παρατήρηση, κυρία Πρόεδρε, αυτό που θα ήθελα να προτείνω και εγώ για τη δική μου έκθεση είναι πριν καταθέσετε τροπολογίες, ρίξτε μια ματιά στην έκθεση, μπείτε στον κόπο να τη διαβάσετε, για να μην υποβάλλετε τροπολογίες που ήδη υπάρχουν στο κείμενό μου. Γιατί τα ακούσαμε αυτά τα επιχειρήματα και είναι πολύ λογικά, τα είδαμε και στην περίπτωση της έκθεσης Βανίστερ Ρόι και Κρέλ. Στην η δική μου έκθεση είναι έτοιμη για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Βέβαια δεν, έχει, δεν υπάρχει ακόμη έτοιμο το έγγραφο. Θα ελεγχθεί τώρα το κείμενο και η αγγλική μετάφραση θα αποσταλεί την Παρασκευή στη Γραμματεία. Την επόμενη εβδομάδα λοιπόν θα λάβετε όλοι το αγγλικό κείμενο της έκθεσης. Οπότε η διορία για τις τροπολογίες είναι ε, τέλη Μαΐου, όπως και για τις υπόλοιπες εκθέσεις. Επαναλαμβάνω, στα τέλη τη εβδομάδα, αρχέ τη επόμενη εβδομάδα, θα λάβετε το αγγλικό κείμενο τη έκθεση. Σε ό,τι αφορά τώρα τη φιλοσοφία του κανονισμού, να δώσω κάποιες ε, εισαγωγικές πληροφορίες για να ξέρουμε όλοι περί τίνος πρόκειται. Τον Ιούλιο αυτό που θα ψηφίσουμε είναι η εντολή προς τους συζητητές για τις διαπραγματεύσεις. Δεν θα είναι τελική ψηφοφορία δηλαδή στην Επιτροπή μας. Απλώς θα είναι ψηφοφορία για τη διαπραγματευτική εντολή προς τους συζητητές. Οπότε στην έκθεσή μου θα περιλάβω και κάποιες προκλητικές παρατηρήσεις προκειμένου να διευρύνω το περιθώριο διαπραγμάτευσης. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν το έχει δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ούτω ή άλλω δεν πρόκειται να δεχτεί τέτοιες προτάσει για πολύ καιρό. Αλλά όλα θα εξαρτηθούν από την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Γιατί χρειαζόμαστε περιθώριο λιγμό στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Θέλουμε να δείξουμε στο Συμβούλιο ότι είμαστε έτοιμοι για διαπραγμάτευση. Ε, και δεν είμαστε μόνο έτοιμοι για την πρώτη ανάγνωση, είμαστε έτοιμοι και για τον τριμερή διάλογο και για τη συνδιαλλαγή και για τη δεύτερη ανάγνωση. Δεν ε, ε, προσβλέπουμε σε ολοκλήρωση του θέματος σε διεκπαιρέωση από την πρώτη ανάγνωση. Προσοχή λοιπόν, υπάρχουν κάποια στοιχεία στην έκθεσή μου που είναι ιδιαίτερα φιλεγόμενα για το Συμβούλιο και προκλητικά. Δεν πρόκειται να διαβάσω όλες τις τροπολογίες, αλλά θα αναφερθώ σε ορισμένα σημεία μόνο. Το ένα αφορά το πεδίο εφαρμογή. Το πιο επίμαχο στοιχείο της έκθεσης είναι ε, η επιλεξιμότητα για την παραγωγική δαπάνη να δοθεί μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ προτείνω να επεκταθεί σε όλες τις επιχειρήσεις. Ε, να φέρεται ειδικό για τις μικρομεσαίες, αλλά να ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις. Λέω λοιπόν στην έκθεσή μου ειδικό για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Κυρίω για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Αυτό σημαίνει όμω και, με τις και για τι υπόλοιπε επιχειρήσει εφόσον συνεργάζονται με τι μικρομεσαίες. Αυτό το σημαίνει ιδιαίτερα σημαντικό για τι εξόχω απόκεντρε περιοχέ. Γιατί εξόχω ε, κέντρες περιοχές ε, ζήτησαν περιορισμό. Είναι πολύ επίμαχο το σημείο. Εγώ θα προσπαθήσω να επιτύχω μία διεύρυνση του πεδίου εφαρμογή για να περιλαμβάνει και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης, θα ζητήσω διαγραφή ενός στοιχείου που είναι ακόμη πιο επίμαχο. Αφορά την απαγόρευση για τι ε, υποδομέ βασικών υπηρεσιών στι πιο αναπτυγμένε περιοχές, ε, μεταφορέ περιβάλλον και πληροφορίες επικοινωνίας. Προτείνω διαγραφή αυτού του σημείου. Και επειδή η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις, γενικές, ε, από τις διάφορες γενικές ειδευθύνσεις είναι επειδή οι ανεπτυγμένες περιοχές τα έχουν ήδη καταφέρει, αυτή είναι η πρώτη απάντηση, ή δεύτερον θα έχουν το Connecting Europe Facility. Αυτά μου λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως ε, η Γενική Διεύθυνση MOVE ε, εξεπλάγει γιατί θεώρησε ότι η απαγόρευση αφορά το Connecting Europe. Δεν φαντάστηκε η, Γενική Διεύθυνση MOVE ότι το Connecting Europe θα χρησιμοποιούνταν ως ε, πρόσχημα για την απαγόρευση στις υποδομές. Οπότε, η λογική ερώτηση είναι ε, αν ε, τα χρήματα πάνε στον οργανισμό θα είναι ακόμη είναι, ταμείο συνοχής ή δεν θα, ισχύει, δεν θα θεωρούνται πια ω ε, τα κονδύλια συνοχή, Γι' αυτό προτείνω σχετική διαγραφή και επίση προτείνω διαγραφή ενό πολύ ενδιαφέροντο ζήτηματο για τον καπνό. Κάποιοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μου είπαν κάτω τα χέρια από τον καπνό. Εγώ παρόλα αυτά θα προτείνω διαγραφή αυτό το σημείο, γιατί είναι ιδεολογικό αυτό το θέμα πώς θα καταπολεμήσουμε το κάπνισμα. Πάντως, το θέμα των υποδομών είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να θετήσουμε μια πολύ σαφή πολιτική θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ή θα ταχθούμε υπέρ ή θα ταχθούμε κατά. Θα πρέπει η θέση μας είναι ξεκάθαρη όμως. Υποδομές και βασικές, για τις βασικές υπηρεσίες, μεταφορά περιβάλλον και τεχνολογίε επικοινωνία και πληροφορία. Νομίζω ότι δεδομένη κρίση θα πρέπει να, είναι ανοιχτό, να ανοιχτό το θέμα. Το ακούσαμε και στην πρωινή συνεδρίαση με του εκπροσώπου των περιφερειακών οργανώσεων. Ένα άλλο θέμα που πολύ δύσκολα θα γίνει δεκτό από το Συμβούλιο, για να μην πω ότι θα απορριφθεί η συλλήφθη, είναι το θέμα των αλλαγών στου θεματικού στόχου. Τρει είναι οι στόχοι που έχουν ε, προταθεί για τη θεματική συγκέντρωση και αναφέρεται και ένα ποσοστό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εδαφική συνεργασία, εκεί έχουμε μια τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Λέει από τους 11 στόχους κρατήστε τους 3. Ενώ στο αναπτυξιακό ταμείο θα πρέπει να, να διαλέξει κανείς 3 στόχους και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα ε, ελαστικότητας. Εγώ προτείνω 4. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος και τέταρτος. Δηλαδή καινοτομία, τεχνολογίες ε, επικοινωνίας και πληροφορίας που αποκλείονται σήμερα, ICT, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενεργειακή αποδοτικότητα. Εγώ προτείνω τρεις λοιπόν στόχους και όχι... Ε, τέσσερις συγγνώμη στόχους και όχι τρεις. Τώρα, ε, σε ό,τι φορά τη στρατηγική, προτείνω όχι 80-20, αλλά 70% για τις πιο αναπτυγμένες περιοχές. Προτείνω μια αλλαγή στα ποσοστά δηλαδή. Και φυσικά κρατάμε το 20% για την ενεργειακή αποδοτικότητα και στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές προτείνω να κατεβούμε από το 50%, να φτάσουμε στο 40% ενδεχομένω. Αυτή είναι η πρόταση και τουλάχιστον 10% για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ε, σημαντικό στοιχείο ιδιαίτερα για την ε, σταδιακή κατάργηση. Είμαι υπέρ της ελαστικότητας, όχι 80 αλλά 70, όχι 20 αλλά 10, όχι 50 συγγνώμη, αλλά 40, δεν αλλάζει η ουσία, το περιεχόμενο, αλλά είμαστε πιο ελαστικοί. Ούτε αλλάζουμε τους θεματικούς στόχους, αλλά διαβρύνουμε το στόχο των επενδύσεων προτεραιότητας. Σε πολλά σημεία προ, προσθέτω και τον πολιτισμό. Ε, την, τον κλάδο του πολιτισμού, τη δημιουργική βιομηχανία. Ο πολιτισμός είναι μια, ένας δημιουργικός κλάδος. Επίσης, προτείνω επιλεξιμότητα για τις υποδομές τουρισμού, πολιτισμού και αθλητισμού. Γιατί έχουμε υποδομές υγείας και εκπαίδευσης. Προτείνω εκτός από την υγεία και την εκπαίδευση τον τουρισμό, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό κατά την ε, έναρξη των διαπραγματεύσεων. Τώρα, ε, δημιουργική βιομηχανία, e-culture και πρόταση για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Προτείνω το θέμα της, ε, της κινητικότητας της πόλης να αλλάξει θέση. Γιατί είναι θέμα χαμηλή χρυσή άνθρακα και προ το παρόν αποκλείεται από τη θεματική συγκέντρωση. Προτείνω να επαναπροσθεθεί στην θεματολογική συγκέντρωση γιατί αφορά τη χαμηλή χρήση άνθρακα. Το urban mobility να μπει στη θεματική συγκέντρωση λοιπόν, η κινητικότητα στι πόλει. Και τα θέματα φυσικά τη ενεργειακή αποδοτικότητα των κτίριων. Τώρα, το θέμα της αντιπαλότητας των πόλεων, ε, η αποκατάσταση των ε, μολυσμένων ε, τόπων, οικοτόπων και ούτω καθεξής. Αυτό προκύπτει από το έγγραφο εργασίας του κοινού στρατηγικού πλαισίου. Χρησιμοποιώ κάποια επιχειρήματα του εγγράφου για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο στις προτεραιότητες για τις επενδύσεις. Επίσης, εκεί που λέμε για τι θαλάσσιες μεταφορές, προτείνω και γενικώ τι μεταφορές, τις πλωτές μεταφορές, όχι μόνο τις θαλάσσιες. Ένα άλλο πολύ επίμαχο στοιχείο είναι η πρόταση για την πλήρη κατάργηση των δικτών από τον κανονισμό. Αυτό φυσικά θα είναι ένα καθόδες στοιχείο της συζήτηση. γιατί και στο έγγραφο αυτό και στο έγγραφο για την εδαφική συνεργασία έχουμε δείκτε των αποτελεσμάτων, ε, του output των νεκρών, όχι των αποτελεσμάτων. Οι δείκτες αποτελεσμάτων θα πρέπει να, να, δημιουργούνται από τη βάση. Ενώ οι δείκτες ε, εκρών ουσιαστικά αφορούν τη συγκέντρωση δεδομένων. Ενδιαφέρον θεμαμένα, αλλά άσχετο με το Αναπτυξιακό Ταμείο, το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προτείνω να μπουν σε εκτελεστικές πράξεις Νομίζω ότι έτσι ενισχύουμε τη δραστηριότητα τη Επιτροπή με τη συμπερίληψη στι εκτελεστικέ πράξει. Αλλιώ θα πρέπει να τροποποιήσουμε. αρχίζουμε τροποποίηση των δικτών και τότε. Τι να σα πω, καλό κουράγιο αν πρέπει να αρχίσουμε να τροποποιούμε του δείκτε. Γιατί μερικοί είναι πολύ, πολύ αμφιλεγόμενοι, πολύ επίμαχοι, άλλοι είναι απλούστατοι, αλλά μερικοί είναι πολύ δύσκολοι. Είναι χρήσιμοι για τη συγκέντρωση δεδομένων, αλλά όχι χρήσιμη για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ούτε για το Ταμείο Συνοχής, ούτε για την Περιφερειακή Συνεργασία. Προτείνω λοιπόν οι δείκτε να μπουν στι εκτελεστικές πράξεις. Σε ό,τι αφορά την αηφόρα ανάπτυξη των πόλεων, το περίφημο 5% που συζητήσαμε και σήμερα στις συμβάσεις. Ας είμαστε ε, συνεπείς. Να είναι και στο γενικό κανονισμό και στο ειδικέ διατάξει για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξη, όπω είπε η Κωνσταντζα. Τα κονδύλια για τις πόλεις δεν είναι περιορισμένα. Μπαίνουν στι επενδύσει ε, προτεραιότητας. Η Επιτροπή προτείνει, και εγώ συμφωνώ, ένα είδο πιλωτικού 5%. Αυτό μπορεί να αφιερωθεί ιδιαίτερο για να δημιουργηθούν ε, οι δεσμοί εταιρικότητα στα δίκτυα μεταξύ των πόλων και των προαστίων. Η πρότασή μου λοιπόν είναι αυτό το 5% να αφιερωθεί στις, στις λειτουργικές αστικές ζώνες. Και ποιες είναι αυτές θα εξαρτηθεί από την σύνταξη της σύμβασης. Στη συμβάση θα πρέπει να έχουμε ένα κατάλογο κριτηρίων που θα γίνονται αποδεκτές σε εθνικό επίπεδο για, τις, για τους λειτουργικούς πόρους, χωρίς νούμερα. Μόνο κριτήρια και να αποφασίζουν οι χώρες τι είδου λειτουργικούς ε, χώρους, λειτουργικέ λειτουργικές ζώνες θέλουν να χρηματοδοτήσουν. Κατά τη γνώμη μου, ε, είναι πόλεις και προάστια. Για να δημιουργήσουμε μια προστιθέμενη αξία, αυτό θα πρέπει να είναι σαφές. Γι' αυτό προτείνω κάτι τέτοιο στις τροπολογίες και επίσης προτείνω διαγραφή, κατάργηση της πλατφόρμας των πόλων, του Urban Platform. Γιατί είναι χρήσιμη η πλατφόρμα αυτή για το πληθυσμιακό στοιχείο, αλλά γνωρίζουμε από ενδιαφερόμενους ότι υπάρχουν ήδη πολλές, πολλοί μηχανισμοί, πολλά μέσα. Αν θέλουν ε, οι οργανώσεις μπορούν να συνεννοηθούν, δεν χρειάζεται η πλατφόρμα των πόλων. Και τι γίνεται με τις περίφημες 300 μεγάλες πόλεις. Ναι, από πολιτική άποψη και για τη συζήτηση καλό ακούγεται για να κινητοποιηθεί ο κόσμος, αλλά είναι κάπως προκλητικό και από άψη έμπρακτη εφαρμογή δεν νομίζω ότι έχει και πολύ νόημα, γι' αυτό προτείνω να καταργηθεί αυτή η πλατφόρμα των πόλων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία, τα πιο επίμαχα από την έκθεσή μου. Επαναλαμβάνω, στα τέλη της τρέχουσα εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης θα λάβετε την πρότασή μου στα αγγλικά πρώτα και θα περιμένω τις αντιδράσεις. Φυσικά θα συναντηθώ με τους σχεδόν ηγητές και θα έχω στενή συνεργασία με τους συνεισηγητές για το γενικό κανονισμό και θέλω να αποφευθούν οπωσδήποτε αντιφάσεις μεταξύ γενικού κανονισμού και ειδικού. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα πολύ γρήγορα οι σχεδόν ηγητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε εδώ είμαι. Κύριε Όρπριχτ, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. των τροπολογιών σας θα γίνει σε συνάντηση με τους σκιώδεις ηγητές πιστεύω αυτήν την εβδομάδα και η βάση είναι αυτά τα οποία πολλές φορές έχουμε επισημάνει σε ανταλλαγές απόψεων. Τα σημεία στα οποία πρέπει να δώσουμε έμφαση. Και θα ήθελα να πω δύο λόγια με τον κίνδυνο να επαναληφθώ Δηλαδή, υποδομές. Στις υποδομές όντως πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις στις υποδομές δεν πρέπει, δεν μπορούν να είναι περιορισμένες σε ορισμένες περιφέρειες μόνο. Πρέπει να είναι στη διάθεση όλων των περιφερειών, ακόμη και των πιο πλούσιων γιατί μπορεί κάπου να υπάρχουν ελλείμματα, φερρυπίν ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών ή ως προς τις νυχτερινές μεταφορές. Το παράδειγμα που αναφέρατε εσείς, ε, το ίντερνετ ε, μεγάλης ταχύτητας, ε, την ευρυζωνική μεταφορά στοιχείων κτλ. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι το θέμα της προαγωγής και υποστήριξης επιχειρήσεων. Δεν θα πρέπει να περιοριζόμαστε μόνο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ανεξαρτήτως μεγέθους θα πρέπει να εξετάζουμε εάν υπάρχει κίνδυνος μετατόπισης απώλειας θέσεων εργασίας δηλαδή. Και αυτό θα το καταθέσουμε με τις τροπολογίες μας. Θεματική ε, συγκέντρωση, θεματολογική συγκέντρωση, Βεβαίω συμφωνούμε με τη βασική αρχή. Θα πρέπει οπωσδήποτε και να ασχοληθούμε με τομείς στους οποίους μπορούμε να προσφέρουμε προσθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά στόχος δεν μπορεί να είναι το 80% κανόνας, δηλαδή για, την, για τις περιφέρειες του στόχου 2, να μείνει ακλόνητος και δίσκαμπτος. Αυτό πρέπει να το συστήσουμε, γιατί υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες ήδη έχουν ολοκληρώσει την ενεργειακή λεγόμενη εξυγίανση κτηρίων, αλλά έχουν μένει πίσω σε άλλα θέματα, σε θέματα φερρυπίν κοινωνικής ενσωμάτωσης, βιώσιμη ή αηφόρου χρήση σπόρων ούτω καθεξής. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε περισσότερη ευελιξία, λιγότερο μονομερή προσέγγιση και να επιδιώξουμε περισσότερο από το περισσότερο προϊόν από αυτό που θα προτείνουμε. Και επίσης, οι δημογραφικές εξελίξεις πιστεύω θα πρέπει να αναφέρονται και σε αυτή την έκθεση ως ουσιαστική τοποθέτηση και όχι παρεπιπτόντως με μία μόνο φράση. Υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες, άλλωστε το έχει η Επισμανική Επιτροπή, έχουν όλο και λιγότερο πληθυσμό, αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα απώλειας κατοίκων και πρέπει και πολιτικά να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Για την προαγωγή του αθλητισμού, του πολιτισμού, του τουρισμού συμφωνούμε απολύτως και θα πρέπει όχι μόνο να δίνονται οι πληροφορίες αλλά και να αναγνωρίσουμε ότι το ε, Ταμείο ήδη από το άρθρο 2 έχει ορίσει αυτούς τους στόχους ως ουσιαστικούς στόχους που εξυπηρετεί. Νομίζω λοιπόν ότι ε, οι προτάσεις με μη, κάποιες μικρές βελτιώσεις μπορούν να, ενσωμα, μπορούν να αποτελέσουν μια έκθεση η οποία θα εγκριθεί από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερο είναι αυτό του καταλόγου 7 που αναφέρατε και εσείς, του περίφημου καταλόγου 7 που πρέπει να απαλληφθεί, δεν μπορεί να παραμείνει. Και πρέπει να επισημάνουμε στο Συμβούλιο ότι υπάρχουν πάντοτε εναλλακτικέ ιδέες, δεν χρειάζεται να βρεθεί κάτι ε, εξ αρχής, υπάρχουν δεδομένες ιδέες. Και επίσης δεν θέλω να επισημάνω εκεί όπου υπάρχουν δυνατότητες για διάθεση κονδυλίων για την ανάπτυξη των αστικών κέντρων από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Θα ήταν καλό να την αναπτύξουν την ε, διαδικασία αυτά τα κράτη και να μην την λησμονούν. Σταματώ εδώ και, και περιμένω τον, ε, την ευκαιρία την Πέμπτη να ε, ψηφίσουμε και ελπίζω με πολύ μεγάλη πλειοψηφία την εκθέση σας. Ευχαριστώ. Κυρία Μάνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω φιλανδικά, εφόσον έχω την δυνατότητα. Ναι. Υπάρχει φιλανδική διερμηνία. Πολύ ωραία. Συνεχίζω λοιπόν στη φιλανδική. Ευχαριστώ το Γιάννη για το εξαιρετικό του έργο, για όλες τις ιδέες που μας ε, υπέβαλε και τις οποίες μπορώ να στηρίξω. Σε ό,τι αφορά τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές, συμφωνώ. Οι πιο ανεπτυγμένες περιοχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από την βοήθεια του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης για τις υποδομές τους. Συμφωνώ με όσο είπε ο Γιάννη. Δεύτερη παρατήρηση. Θα πρέπει το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης να είναι πιο ευέλικτο για τα μεγάλα ζητηγικά θέματα. Αυτό είναι δικαιολογημένο. Το σχολιάζω και εγώ στην έκθεσή μου και σωστά το επισημαίνει και ο Γιάννη. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες θα συμφωνήσω απολύτως. Η άποψη του Γιάννη είναι πολύ σωστή. Για την εδαφική συνεργασία, για το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ναι, να διαγραφούν. Και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Το αναφέρω και εγώ στην έκθεσή μου για την εδαφική συνεργασία, σε ό,τι αφορά τα αστικά κέντρα. Ε, και εδώ θα συμφωνήσω. Ουδέποτε ήμουν υπέρ αυτής, αυτού του καταλόγου, ενό σταθερού καταλόγου πόλεων ή των αστικών πλατφορμών, όπω ονομάζεται για τη στιγμή. Όχι, θα πρέπει να ορίσουμε προποθέσει ανάλογα με τι ανάγκε τη κάθε χώρα. και θα συμφωνήσω απολύτως με όσα υπόθηκαν για τι ε, ζώνε των αστικών κέντρων. Νομίζω υπάρχει μεγάλη σύγκληση μεταξύ των εκθέσεών μα στο σημείο αυτό. Μόλι λάβουμε το κείμενο και στη μετάφραση θα τα μελετήσουμε με ακόμη μεγαλύτερη προσοχή, αλλά άκουσα τώρα μου φαίνονται εξαιρετικά. Ευχαριστώ από ό,τι καταλαβαίνω κυρία Ντελή, δεν εδώ. Κύριος Γκλάφικ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερο τον Γιάννη που δείχνει τέτοιο ενθουσιασμό στην εκπόνηση αυτή τη έκθεσης. Συμφωνώ με τις προτάσεις του. Και έχω σημειώσει όλα τα σχόλια που ακούστηκαν. Οι μεγάλες εταιρείες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και οι μεγάλες όμως επιχειρήσεις πολλά επενδύουν στην κοινοτομία και την έρευνα να τις ε, σκεφτούμε και αυτές, γιατί μιλούμε μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, δηλαδή να, να καλυφθούν ο τουρισμός, η βιομηχανία, ο κλάδος της δημιουργίας και ο, αθλη, και ο αθλητισμός. Και αυτό είναι πολύ καλή ιδέα. Και τελευταίο σχόλιο για τις πιο αναπτυγμένες περιοχές. Η αστική κινητικότητα και βιώσιμε μεταφορέ βεβαίω είναι θεμετή στόχη. Επιφυλάσσομαι για τι μελλοντικέ μα συζητήσει. Κυρία Ένστ. Ε, είχε έτσι, Η σειρά μου δεν είναι. Κυρία Ένστ. Ναι, πρόεδρε, συγγνώμη, δεν σας είχα καταλάβει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τους δύο συγγητές. Τον εισηγητή, ε, πολλά είναι τα θέματα που μπορούμε να υποστηρίξουμε εδώ. Δεν είναι βέβαια όλα ε, επαναστατικέ προτάσει. Θα έχουμε ξαναδεί στην Επιτροπή των Περιφερειών, αλλά εν πάση περιπτώσει μα αρέσουν και υποστηρίζουμε βεβαίω και την απέτηση όχι για τι μικρομεσαίε, αλλά κυρίω για τι μικρομεσαίε. Δηλαδή το ότι δεν είναι αποκλειστικά, αλλά κατά κύριο λόγο μικρομεσαίε επιχειρήσει στο μα, μα αρέσει πάρα πολύ. Ε, στο θέμα των υποδομών στις ε, πόλεις, στα αστικά κέντρα βεβαίως, ναι, είμαστε ευχαριστημένοι και το έχουμε συστήσει πολλέ φορές. Νομίζω ότι θα είχε νόημα να συζητήσουμε διάφορα θέματα τα οποία ίσως να έχουν κάποιες δυσκολίες. Για τα νούμερα 3 ή 4 δεν ξέρω πόσο επαναστατικό μπορεί να είναι. Δεν είμαι βεβαία δηλαδή ότι αρκεί στην η θεματική συγκέντρωση με την πρόταση αυτή που έχετε για να υλοποιηθεί. Τα ποσοστά 70 κτλ. Ίσως θα πρέπει να το συστήσουμε στις συνεδρίες των σκιωδών. Ίσως να αρκεί, ίσως χρειάζεται λίγο τη δουλειά. Βεβαίως υποστηρίζουμε τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον τουρισμό. Πρόταση της Επιτροπής Πολιτισμού άλλωστε. Διάσταση των αστικών κέντρων. Θα ήθελα εδώ να ρωτήσω εάν η πρόταση της Επιτροπής των Περιφερειών είναι βάση ή την έχετε υπόψη σας, σε πάση περιπτώσει, διατύπωση των ε, προτάσεών σας, εάν σας έχει απασχολήσει, γιατί είναι θέμα και αρμοδιότητα τη Επιτροπή των Περιφερειών, θα μπορούσα να μιλήσει για ανάπτυξη αστικών κέντρων κλπ. Το είχατε αυτό υπόψη ή θέλετε να συστήσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο προκειμένου. Ο κατάλογος των κριτηρίων από το γενικό κανονισμό πιστεύω μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση και κατά τα άλλα Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά καλά και περιμένω να τα συστήσουμε και στους, στις συνεδρίες των σκιωδών. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ε, πολύ έχουν ζήσει τον λόγο. Ως το δυνατόν πιο σύντομα, Μαρία Τερέση Σάντσι Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω να έρθω στο στον Γιάννη για τη δουλειά του και για τις πολύ συγκεκριμένε προτάσεις. Ε, βεβαίως, Τρέφουμε κάθε ψήφινο στο πρόσωπό του για να βελτιώσει το κανονισμό αυτών. Τέσσερα είναι τα σημαντικά για μας σημεία. Η αιρεσιμότητα των σχεδίων υποδομών για τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές, ε, συγκέντρωση θεματολογική για τις ε, περιφέρειες σε μετάβαση, μικροεπιχειρήσεις, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολιτισμός και κλάδος του πολιτισμού, στις επενδύσεις, που ξέρετε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα Ο πολιτισμός και ο χώρος της δημιουργίας αποτελεί το 4,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ με 5 εκατομμύρια απασχολούμενους. Ο κλάδος του πολιτισμού και της δημιουργίας βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη στην Ευρώπη και πρέπει εξάπαντος να υπαχθεί στα άρθρα 3 και 5. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιάν. Δεν ξέρω πώς να χαρακτηρίσω την προσέγγιση του υψηλής ποιότητας, άμεση κτλ. Είσαι πολύ, πολύ καλός, πολύ δυνατός. Μπορεί να μην κέρδισετε αγώνες αποδοσφαιρικούς, ε, αλλά πάντως βλέπω ότι είσαι στη θέση αυτή πολύ ε, αποτελεσματικός. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει στη δική μας την περίπτωση με την Κωνσταντς τώρα ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί με πιο συγκεκριμένου όρου η πρόταση. Και θα ήθελα ένα συγκεκριμένο σημείο να υπογραμμίσω το 10% με την τροπολογία που ορίζει ότι μέχρι 10% από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να δαπανηθεί έξω από την εδαφική περιφέρεια ε, Βλέπουμε όμως ότι σχεδόν ποτέ δεν γίνεται αυτή η δαπάνη, ποτέ δεν ξεφεύγουμε δηλαδή από τα όρια τα εδαφικά. Ε, αν όμως θέλουμε να αναπτύξουμε ένα νέο πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, αν θέλουμε να έχουμε περισσότερη αποτελεσματικότητα στην ε, συνεργασία και τις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, μεταξύ αστικών κέντρων, δηλαδή μεταξύ όλων αυτών οι οποίοι πράγματι δραστηριοποιούνται και ε, έχουν πάρει το δρόμο της ε, αριστείας, δεν ε, πρέπει να τους ε, φράσουμε το δρόμο αυτό, χωρίς να θέλουμε βεβαίως να υποχρεώσουμε κανέναν. Τους καλούμε όλους να βρούνε τέρους, να αναπτύξουν προς προτεραιότητες, ε, σχέσεις, φερειπίν στο χώρο της γνώσης και όλα αυτά τα πράγματα. Εάν θέλετε να συνεργαστείτε, τα κέντρα αριστείας βοηθούν γι' αυτό. Μπορεί κανείς να διδαχθεί τι σημαίνει ε, συνεργασία. Σήμερα είχαμε ένα, δείπνο, ένα γεύμα μάλλον συνεργασίας για το χώρο της ε, φαρμακευτικής βιομηχανίας ε, και τα λοιπά και της έρευνας. Πολύ ωραίο το φαγητό. λοιπόν ρώτησα κάποιους από πού είστε εσείς. Α, μου λένε από την Ανατολική Ευρώπη. Και λέω ότι έτσι γίνεται. έτσι γίνεται μου λένε. Δηλαδή εάν δεν δαπανούμε χρήματα για τις, ψη... για τις πλούσιες περιοχές που θα τις οθήσουμε με τον τρόπο αυτό να συνεργαστούν με τις φτωχότερες αλλά και για τις φτωχότερες για να αναζητήσουν εταίρους, τότε το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Χρειάζεται δηλαδή άλλος τρόπος να προσεγγίσουμε τον εταίρο, άλλο τρόπο, άλλος τρόπος να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις εταιρικέ σχέσεις. Πρέπει να συνεργαζόμαστε περισσότερο για την περιφερειακή ανάπτυξη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όπως θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Επιτροπή για την, για την ε, υλοποίηση του στόχου της Ευρώπης 2020 και δεν θα ήθελα ε, να προσθέσω εδώ μια ερώτηση, αυτό το ποσοστιαίο που αναφέρεται. Ίσως να μπορεί να αποτελέσει ένα νέο χώρο συνεργασίας στην Ευρώπη. Γι' αυτό το 1% που προτείνω εγώ, όχι μόνο γραφειοκρατία, αλλά απλώς μία όθηση, ένα κίνητρο για να κοιτάμε και κάπου αλλού. Θα ήθελα να επισημάνω, λέει η κυρία Πρόεδρος, ότι όσο έτρωγε αυτό το υπέροχο γεύμα ο Λάμπερτ, εμείς μας με την κυρία Σρότερ και άλλους είχαμε συνάντηση με άτομα με αναπηρίες, όπου δεν προσφερόταν το δείπνο. Αυτό, το οποίο, αυτό που λέω είναι ότι πρέπει κανείς να προσέχει τι διαλέγει για το μεσημεριανό του, γιατί εμείς μαθάμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα Κύριε Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Ε, συμφωνώ με τον ε, συγκητή ότι πρέπει να ε, διαγραφεί το, το σημείο εκείνο στο κεφάλαιο 3 που αναφέρει ότι οι αναπτυγμένες περιοχές δεν πρέπει να χρηματοδοτούνται για επενδύσεις στο περιβάλλον και στις μεταφορές. Θα έλεγα αντίθετα θα πρέπει να ευνοηθούν οι καινοτόμες επενδύσεις, ιδιαίτερα οι πράσινες επενδύσεις, τόσο σε θέματα μεταφορών όσο και στα θέματα των υπηρεσιών των οικοστημάτων. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε ακόμα και στι αναπτυγμένε περιοχέ είναι ο μετασχηματισμό του και η εξέλιξή του σε πιο πράσινε κατευθύνσει και πιο βιώσιμε κατευθύνσει. Αλλιώ τι παγιδεύουμε σε συντήρηση παλιών υποδομών. Ε, το δεύτερο που θα ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι σε σχέση με του κλιματικού στόχου και με την εξοικονόμηση ενέργεια και τι ανώσιμε πηγέ, σαν πράσινοι προτείνουμε να αυξηθεί το ποσοστό από 20% 25% για τη χρηματοδότηση κλιματικών στόχων για τις πιο αναπτυγμένες και τις μεταβατικές περιφέρειες και για τις λιγότερο αναπτυγμένες από το ποσοστό του 6% στο 15% σαν ε, στόχους. Ε, πιστεύω ε, ότι είναι πολύ σημαντικό να χρηματοδοτηθούν και παρεμβάσει στον πολιτισμό, γιατί ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία ο πολιτισμός είναι και στοιχείο της περιφερειακής ανάπτυξης. Δεν έχει μόνο αξία ω ίδιο, ω ίδια δραστηριότητα, πολιτική δραστηριότητα, αλλά και πολύ μεγάλη σημασία και μπορεί να δημιουργήσει πολλέ θέσει εργασία σε περιφερειακό επίπεδο, ιδιαίτερα μέσα από την πολιτιστική δράση. Θα, θα συμφωνούσα ότι πρέπει να ενισχυθούν ε, όχι μόνο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και οι κοινωνικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις μέσα από το Ταμείο. Είναι κάτι που ε, πολλές φορές το ξεχνάμε, άρα πρέπει να δούμε και τέτοιες συνεργασίες με κοινωνικές συνεταιριστικέ επιχειρήσει. Ε, θα έλεγα ότι πράγματι συμφωνούμε να μην υπάρχει εξαντλητικό κατάλογος των πόλεων, αλλά κριτήρια για τα, τη συμμετοχή των πόλεων στα προγράμματα, ιδιαίτερα κριτήρια που να αναβαθμίσουν και περιοχές που αντιμετωπίζουν κρίση σήμερα μέσα στις πόλεις. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχει επίση ανάγκη νομίζω να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην κινητικότητα και στην υπεθρό αλλά χωρί να ξεχνάμε τα νησιά. Θα ήθελα, επειδή κατάγομαι και από μια νησιωτική περιφέρεια, να πω ότι αν μιλάμε για αυτοκινητοδρόμου και σιδηρόδρομο για την υπηρετική Ευρώπη, τα νησιά έχουν τη θάλασσα, αλλά αν δεν υπάρχει υποδομή που είναι τα πλοία, δεν υπάρχει σύνδεση. Και αυτό κινδυνεύουμε πολλέ φορέ να το πάθουμε στι νησιωτικέ περιοχέ στην Ελλάδα, δηλαδή να μείνουμε χωρί πλοία. Τα πλοία είναι υποδομή γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Πολύ σπάνια υπάρχει το αεροπλάνο, αλλά και αυτό δεν μπορεί να είναι λύση για όλους. Άρα λοιπόν οι υποδομές είναι πλοία για την κινητικότητα και πολύ περισσότερο για τη βιώσιμη κινητικότητα στα νησιά, αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα καλό εργαλείο το Περιφερειακό Ταμείο για να αλλάξουμε και την αυτιλία, να γίνει πιο πράσινη αυτιλία. Αφού έχουμε ένα σύνολο ε, νομοθεσιών που βάζουν πιο υψηλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τα πλοία, είναι ευκαιρία να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις αλλαγές σε ένα κάποιο βαθμό ή να ενθαρρύνουμε αν θέλετε αυτές τις αλλαγέ, έτσι ώστε πράγματι να Έχουμε υποδομές και για την ε, νησιωτική χώρα, νησιωτικές περιοχές, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πιο πράσινες υποδομές για αυτές τις περιοχές. Και, α, και θέλω, ήθελα να πω που, κάτι που στάμε συνέχεια, οι δείκτες. Ανεξάρτητα που θα μπουν οι διάφοροι δείκτες, πρέπει να μπορούν να περιγράψουν αυτό που θα θέλαμε. Αυτό που λέμε αηφορία, αυτό που λέμε κοινωνική συνοχή, ε, πραγματική ευημερία, βιώσιμη ευημερία. Αυτό πρέπει να περιγράφουν οι δείκτες και να μην είναι απλώς στατικοί δείκτες μερικά χιλιόμετρα ή πόσο απορροφήθηκαν οι πόροι ή πόσοι άνθρωποι εξυπηρετούνται, αλλά αν πραγματικά εξυπηρετούνται και αν πράγματι επιτυγχάνουν τη στόχη του Ευρώπη 2020. Thank you uh, very much. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι εξαντλούμε τον κατάλογο των αγορητών και ρωτώ εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μπορέσει να συνέλθει από το σοκ και να πάρει μια ανάσα για να απαντήσει. Ναι, βεβαίω, βεβαίω, ε, εισαγωγή δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Πάρα μόνο ότι ίσω να απογοητευτούν οι πάντες αν χρειαστεί. Εν πάση περιπτώσει, ε, έχω απαντήσει νομίζω Μάλλον, εάν χρειαστεί να απαντήσω σε όλα τα σημεία, μάλλον θα σα κρατήσω πάρα πολύ ώρα, γι' αυτό θα επικεντρωθώ σε ορισμένα. Και θα ήταν καλό, νομίζω, να αντιληφθούμε περισσότερο τι εννοεί ο, ο εισηγητή ε, με τον όρο μεγάλε επιχειρήσει. Τι εννοεί ο Μήλου, εννοεί μεγαλύτερε επιχειρήσει. Είναι κάτι το οποίο μα είχε απασχολήσει βεβαίω στο πλαίσιο τη ε, έρευνά μα. Ε, αν και το να ανοίξουμε τις δυνατότητες και για τις πραγματικά μεγάλες επιχειρήσεις δεν είναι μια καλή λύση από ό,τι εκτιμούμε. Ε, για το θέμα λοιπόν των υποδομών, βλέπω ότι πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να διευκρινιστεί και να αφήσουμε κατά μέρο στο στόχο αυτόν της ε, γενικεύσεις. Ε, βεβαίως οι υποδομές μπορούν να δραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο, αλλά πιο σημαντικό είναι τι είδους κλίμακα και τι τύπο ε, έργων θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε όχι αυτοκινητοδρόμους και όχι ε, μονάδες διαχείρισης αποβλήτων γιατί εκεί έχουμε τις δυνατότητες της ανάπτυξης του δυναμικού της κοινοτομίας σε αυτές τις περιφέρειες. Το θέμα των καπνών είναι ζήτημα πολιτικής συνοχής, μάλλον συν, ε, πολιτικής συνέπειας. Έχουμε λάβει αποφάσεις για την σταδιακή κατάργηση και απαγόρευση της ε, διαφήμισης καπνού, της απαγορεύσης του καπνίσματος σε κλειστούς χώρους, της απαγορεύσης της χορηγίας προϊόντων καπνού σε αθλητικές εκδηλώσεις. Επομένως, πρέπει να αποστείλουμε ένα μήνυμα συνεπέ με όλη αυτή την πολιτική. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε, όπω λέτε, σε ένα θετικό μήνυμα ότι η Επιτροπή σα θέλει να υποστηρίξει τον καπνό, τα προϊόντα καπνού. Και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ένα σημείο, χωρί να θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε, γιατί ξέρω ότι θα, έχουμε ότι θα έχουμε στο μέλλον περισσότερο χρόνο για να το συζητήσουμε. Το επίπεδο των φιλοδοξιών που ενδεχομένω τρέφουμε για το 70 και το 40. Γιατί μας ε, ε, ενδιαφέρει, διότι όταν συνδυαστούμε συνδυάσουμε με άλλες προτάσεις, ICT δηλαδή, κυρίως με τις πληροφορίες, έχουμε τελείως διαφορετικές ε, φιλοδοξίες και φαίνεται σαν να λέμε ότι ενώ χρειάζεται περισσότερη καινοτομία, περισσότερη ανάπτυξη και ιδιαίτερα σε ορισμένες περιοχές, περιφέρειες πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση, φαίνεται να συμπεριφερόμαστε να μην έχει υπάρξει κανένα πρόβλημα και να βαίνουν τα πράγματα ομαλώς. Για το περιεχόμενο νομίζω ότι μπορούμε να συστήσουμε με τον εισηγητή τις διαφορετικές επιλογές. Βλέπουμε ότι και ο κανονισμός μπορεί να αποτελέσει ένα πρόσφορο μέσον, αλλά και η κατεξουσιοδότηση πράξη. Ε, στο θέμα των αστικών κέντρων, από ό,τι έχουμε αντιληφθεί από τα όσα μας είπε ο εισηγητής, ο στόχος του είναι μάλλον να διευκρινίσει και όχι να αλλάξει άρδιν τις προτάσεις της Επιτροπής και ως τούτου το αντιλαμβανόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Μια αστική πλατφόρμα ε, μπορεί να διαδραματίσει έναν ρόλο ενδιαφέροντα, αλλά θα θέλαμε σε συνεργασία με τον εισηγητή να αντιληφθούμε ακριβώ τι εννοεί και ποιο μπορεί να είναι αυτό ο ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Γιάννη, θε να σχολιάσει τίποτα. Ευχαριστώ καταρχήν για τι παρατηρήσει σα, που ήταν γενικώ ε, θετικέ. Και σα ευχαριστώ για την κατανόηση που δείξατε ε, πιστεύω ότι εστερνιζόμαστε πολλές απόψεις. Περιμένω πάντως με ανυπομονησία και τις τροπολογίες σας. Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Περιφερειών, από την αρχή συνεργάστηκα με την Επιτροπή Περιφερειών. Μπορείτε, μπορούμε να συζητάμε ποιος ήταν ο πρώτος. Πάντως, ε, οι εισηγητές ε, έχουν παρόμοια προσέγγιση. Μερικέ φορέ. η Επιτροπή Περιφερειών ήταν πιο ριζοσπαστή και μερικέ φορέ εγώ. Πάντως γενικώ είμαστε στην ίδια γραμμή πλέψη. Τώρα, τα κριτήρια για του λειτουργικού χώρου, δεν θα πρέπει να, να υποβάλλονται άνωθεν από τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να τα επεξεργάζονται αυτά τα κράτη-μέλη τα κριτήρια, να μην επιβάλλονται από, κεντρικά από τις Βρυξέλλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πρόταση του Λάμπερτ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το συζητήσουμε με ενδιαφέρον. Για τους δείκτες. Όπως είπε ο συνάδελφος εγώ, ε, το θέμα είναι ε, δεν μπορεί οι δείκτες να ε, καταρτίζονται από τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να ξεκινούν από τη βάση. Τα αποτελέσματα μπορούμε να κρίνουμε. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό το σημείο για τους δείκτες. Να βγουν στις εκτελεστικές πράξεις είναι πιο σωστή εκεί η συμπερίληψη. Πιστεύω ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη σύγκληση και θα πρέπει να διευκρινιστεί η κατάσταση. Το πιο δύσκολο πάντως, καταρχήν, το γενικό πολιτικό μήνυμα, Πίτερ, θα ήθελα να πω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι θα πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στους τοπικούς παράγοντες στους περιφερειακούς φορείς είναι λογική. Δεν μπορούμε όλα να τα αποφασίζουμε στις Βρυξέλλες. Δεν μπορούμε εμείς να υπαγορεύουμε στις τοπικές και περιφερειακές αρχές τι θα κάνουν. Να τους πούμε αυτές οι υποδομές, να, σε αυτές οι υποδομές να Είναι λογική οι τοπικοί και περιφερειακή περιφερειακοί παράγοντες. Ξέρουν τι χρειάζονται. Να μην τους αντιμετωπίζουμε σαν μωρά παιδιά και να τους επιβάλλουμε τα πάντα, να αποφασίζουμε εμείς για τα πάντα. Αυτό το πρόβλημα ισχύει για τις συμβάσεις, για, τις, ε, για τα επιχειρησιακά προγράμματα, για τις διαπραγματεύσεις με τις ε, περιφέρειες, να μην τις αποκλείουμε. Από την αρχή να τις ε, συμπεριλαμβάνουμε. Σε ό,τι αφορά το καπνό. Είναι λογικό, δεν είναι αυτό το θέμα, είναι λογικό ή όχι. Το θέμα είναι να είναι σωστή αυτό το, το σημείο για να το συμπεριλάβουμε. Θα πρέπει στο ΦΕΔΕ να περιλάβουμε ότι δεν, μπορούμε να χρημα... ότι δεν θα, πρέπει... ότι θα πρέπει να χρηματοδοτούμε στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλά που δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούμε. Γιατί να λέμε τον καπνό, σαν και καλά. Δεν είμαι, δεν είμαι κατά του καπνού. Συ... Ζητάμε για τι υποδομέ, για την καινοτομία, για τι τεχνολογίε πληροφορίε, επικοινωνία και... και τον καπνό. Από πού και ω πού. Δεν είμαι κατά. Δεν... Απλώς είναι άσκοπο το σημείο αυτό, είναι ακατάλληλο αυτό το σημείο. Τώρα, τα ποσοστά 80%, 70% δεν είναι θέμα φιλοδοξία, είναι θέμα ελαστικότητας. Θέλουμε περισσότερη ελαστικότητα, ναι ή όχι. Το 80% είναι πολύ αυστηρό κατά τη γνώμη μου. Μπορούμε να συζητήσουμε το επίπεδο ή να μην έχουμε τρεις αλλά τέσσερις θεματικούς στόχους. Αυτή είναι η ελαστικότητα. Αυτό επιδιώκουμε. Και κάτι που αναφέρθηκε και προηγουμένως. Δύο στοιχεία για την ακρίβεια που δεν ανέφερα εγώ, τα ξέχασα. Το ένα αφορά την εκχώρηση της διαχείρισης των ταμείων στο επίπεδο των πόλεων. Ένας από τους σημαντικούς στόχους. Το επίπεδο εκχώρησης θα είναι επίμαχο για πολλά κράτη-μέλη. Πάντως η εκχώρηση προς τις πόλεις είναι κέριο σημείο και καινούριο, καινοτόμο. Δίνουμε μάχη εδώ και χρόνια γι' αυτό. Άλλο σημείο είναι τα, η κλίμακα της αριστείας εν του 2020. Θα περιληφθεί στο ΦΕΝΤΕΡ. Θα γίνει μια διασύνδεση του ΦΕΝΤΕΡ με τον ορίζοντα το 2020. Κάτι άλλο που δεν συζητήσαμε αφορά την πραγματική συγκέντρωση και την έλλειψη ελαστικότητας. Είναι η απόφαση για το ESF και τα αυστηρά κονδύλια του, του Κοινωνικού Ταμείου. 27% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες κτλ. Αυτά τα ποσοστά είναι αναλεστικά, απαράδεκτα. Αλλά δεν είναι δικό μας πρόβλημα αυτό. Είναι μια συμφωνία που έγινε μεταξύ των κρατών μελών και θα είναι πολύ δύσκολο να την αλλάξουμε. Θα πρέπει όμως να έχουμε στενή συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης, ώστε τουλάχιστον το πεδίο εφαρμογή να διευρυνθεί του Κοινωνικού Ταμείου. Γιατί στην Πολωνία έχουμε τώρα 12%. Ε, θα αυξηθεί στο 27%. 100% αύξηση δηλαδή. Το θέμα είναι να χρησιμοποιηθεί με λογικό τρόπο. Δεν το ανέφερα, γιατί δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογή του δικού μου κανονισμού, του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ευχαριστώ, θα το συζητήσω με τους σκιώδης ηγητές. Πάντως πιστεύω ότι υπάρχει σύμπνοια και ευελπιστώ ότι θα βρεθούν συμβαστικέ λύσει και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Ευχαριστώ, Γιάννη. Η προθεσμία για τι τροπολογίε λήγει στι 31 Μαου στι 6 το απόγευμα. Θα προσπαθήσουμε να ολοκληρώσουμε τις μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες το συντομότερο δυνατό και να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη ημέρης διάταξη, έκθεση Ρίκα Μάνερ. Βρισκόμαστε σε μια τραγική κατάσταση ως προς το χρονοδιάγραμμα. Ο χρόνος μας πιέζει, έχουμε μείνει πολύ πίσω, γι' αυτό παρακαλώ θερμά να είστε λακωνικότατοι. Άλλωστε είναι θέμα που το έχουμε συζητήσει πολλά και. Ρίκα, έχει το λόγο. But after no? After ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. και να ομαδοποιήσω τα διαφορετικά στοιχεία της ε, παρέμβασης μου. Θα έχετε δει τις ε, πρώτες τροπολογίες που έχω υποβάλει. Δεν θέλω να επανέλθω στην κάθε μια από αυτές, διότι τις έχουμε ήδη συζητήσει. Και μάλιστα δύο φορές. Δεύτερο, δεύτερη παρτίδα των τροπολογιών που κατατέθηκαν και σε αυτές θέλω και να σταθώ. Έχουμε μια πρώτη ομάδα τροπολογιών που αφορούν τα δημοσιονομικά, το 7%, την ευελιξία μεταξύ των διαφορών κεφαλαίων, το 15% την θεματική συγκέντρωση, στοιχεία που είχα ήδη αναφέρει σε προηγούμενες συνεδριάσεις. Ευελιξία και για τη θεματική συγκέντρωση, προτεραιότητες της επενδύσεις. Εδώ έχω διευρύνει κάπως τον κατάλογο προτεραιοτήτων. Στο κείμενο για την εδαφική συνεργασία στην Ευρώπη. Γίνεται λόγος πια και για τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν οι υποδομές. Αυτά για την πρώτη ομάδα των τροπολογιών. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες Αυτέ που θα υποβληθούν στο τέλο του μήνα. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο θέλω να σχολιάσω, είναι πολύ σημαντικό. Το συζητήσαμε και στι συναντήσει με του σκιώδους, συζητητέ τη μακρο Θεωρούμε ότι οι μακροπεριφέρειες έχουν ιδιαίτερη σημασία. Και μας ενδιαφέρει μέσω των μηχανισμών της περιφερειακής ανάπτυξης χωρίς να δημιουργούνται νέα χρηματοδοτικά μέσα για τις μακροπεριφέρειες, να τις στηρίξουμε. Νομίζω ότι συμφωνούμε για το γεγονός ότι οι μακροπεριφέρειες θα πρέπει να στηρίζονται μέσω διαφορετικών διάβλων. Δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με ε, περιφερειακή συνεργασία. Εδώ θα πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια αυτή τη έννοια όπω την αντιλαμβανόμαστε ω τώρα. Έχουμε πάει ως τώρα καλά στην... στο τμήμα του κειμένου που αφορά τι μακροπεριφέρειες. Μπορούμε πάντοτε να επιφέρουμε με βελτιώσεις με κάποιε τροπολογίε και νομίζω ότι εδώ υπάρχει και συνενέση μεταξύ των διαφορών πολιτικών ομάδων. Για του δείκτε τώρα, όπω είχα πει και προηγουμένως, θα προτείνω για την εδαφική συνεργασία να εγκαταλείψουμε το σύστημα των δικτών εδώ δεν εξυπηρετούν τους στόχου των διαφορών ε, τρεχόντων προγραμμάτων. Το ίδιο και για το ΦΕΝΤΕΡ, το Ταμείο περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό που συζητήσαμε από το προηγούμενο σημείο της σημερινή διάταξη. δεν ε, προσφέρουν καμία σαφήνεια οι δείκτε. Ως προς την ευελιξία, στο άρθρο 7, Ιδίω για το Ταμείο Περιφερειακή ανάπτυξη. εδώ θα ήθελα να πετύχουμε μεγαλύτερη ευελιξία ώστε να μπορούμε να, να τα βάλουμε εύκολα τις προτεραιότητες τις επενδυτικές. Ανάλογα με τα θέματα δηλαδή που προτείνονται να μπορούμε και να επιλέξουμε. Συχνά ένα θέμα πρέπει να επιλογεί, να επιλεγεί θέμα που πηγαίνει παράλληλα και με τις επενδυτικές μας προτεραιότητες. Εδώ χρειάζεται λοιπόν διαλλακτικότητα. Αυτό αναφέρθηκε και στο επίπεδο των κοινών διατάξεων, όπω ή άλλω. Οι γενικέ λοιπόν γραμμέ έχω την εντύπωση ότι το κείμενο για την εδαφική συνεργασία στην Ευρώπη θα μα επιτρέψει να επιτελέσουμε πρόοδο στο όλο θέμα. Δεν θέλουμε να εξουθολογήσουμε υπερβολικά τα πράγματα σε σχέση με τι κοινέ διατάξει στο κείμενο για το Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, απλώ να σεβαστούμε τι διάφορε ιδιαίτερε ανάγκε ίσως να χρειαστεί να υπάρξει και μια αναθεώρηση. Ενδιάμεση αναθεώρηση κατά τη διάρκεια ζωή των διαφορών προγραμμάτων και θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά. Αυτά ήταν σύντομα τα σχόλια που ήθελα εγώ να κάνω. Θα υποβάλλουμε πλέον τροπολογίες για τα θέματα αυτά στο τέλο του Μαΐου και θα συνεχίσουμε να συζητούμε ενεργά με τους διάφορους κοιόδους εισηγητές ε, τα διάφορα κεντρικά σημεία. Θα ήθελα τώρα τα σχόλιά σας. Είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό και βεβαίω θα είμαι και σε επαφή με του εκπροσώπου τη Επιτροπή των Περιφερειών που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Διάβασα το κείμενό του, ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικό, πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο και θα ήθελα να έχω και τι δικέ του απόψει για την εδαφική συνεργασία. Ευχαριστώ να καλέσω τον ε, συνάδελφο από την Επιτροπή των Περιφερειών, τον κύριο Όσφαλτ, να μα παρουσιάσει τη δική του τοποθέτηση. Ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε την δυνατότητα για συνεργασία αυτή τη φορά ε, με την Επιτροπή, με την Επιτροπή των Περιφερειών, Συναντιόμαστε βεβαίως στις ε, open days, ε, μέρες ανοιχτές στο κοινό, αλλά ε, δεν μπορούμε πάντοτε να διαπιστώνουμε σημεία συμφωνίας με πιο ενδελεχή συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το θέμα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι δεν έχει ακόμα κλείσει το θέμα της συζήτησης και άρα μπορεί μέχρι την Παρασκευή να βρούμε μία λύση. Βεβαίως χαιρόμαστε που υπάρχει συγκεκριμένο κανονισμός. Σημαντικό είναι ότι υπάρχει κανονισμός για τα μικρότερα προγράμματα συνεργασίας πέραν των συνόρων η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει εάν μπορεί να εφαρμόσει τα μέτρα αμέσως ως μέσα στα, μικρά προγράμματα, στα προγράμματα συνεργασίας πέραν των συνόρων, τα μικρότερα σε σχέση με τα μεγαλύτερα, για να μην χάσουμε καθόλου ε, από την αποτελεσματικότητά μας. Επίσης θα, προσπαθήσουμε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε και τριμερή συνεργασία μεταξύ χωρών ε, γειτονικών η οποία θα ε, ενίσχυε και την ακαιρεότητα των προγραμμάτων αυτών. Νομίζω ότι η διασυνοριακή συνεργασία θα πρέπει ιδιαίτερα να επιδιώκει όχι μόνο η αυτόματα την αρχή της θεματικής συγκέντρωσης, αλλά να επιδιώκει να ενισχύσει την ε, ε, αίσθηση του ανήκει στην Ευρώπη και στόχους της Ευρώπης του 2020 που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν σε διαφορετικό επίπεδο τόσο ικανοποιητικά. Επίσης, σε διασυνοριακό επίπεδο, πιστεύω ότι η θεματική συγκέντρωση και κυρίως η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί ή πρέπει να επιδιώκει βεβαίως κατά κύριο λόγο την ε, ε, στρατηγική του 2020, αλλά πάνω από όλα να προτείνει προτάσεις ε, ή συνθήκες για την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή. Δηλαδή, εάν εφαρμόσουμε έρευνα και ανάπτυξη. Υπάρχουν τομείς όπου θα πρέπει να προσδορίσουμε άλλες προτεραιότητες, συνθήκες για ευρωπαϊκή ανάπτυξη και επίσης στη σύγχρηματοδότηση, στο επίπεδο της σύγχρηματοδότησης θα πρέπει πιστεύω να τηρηθούν οι κανόνες που έχουν ισχύσει μέχρι τώρα αρχές από το Γενικό Κανονισμό, δηλαδή να διαφυλαχθεί το αυτό επίπεδο συγχρηματοδότησης, κυρίως για την ανάπτυξη και της εργασίας, για όλες τις περιφέρειες. Θα πρέπει να έχουν δηλαδή όλες το ίδιο επίπεδο συγχρηματοδότησης. Το ίδιο θα ήθελα να αναφέρω και για τον συντονισμό των κονδυλίων. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε τον συντονισμό των κονδυλίων, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά σε, και σε εθνικό επίπεδο, να καλέσουμε εκείνους οι οποίοι διαχειρίζονται τα σχέδια αυτά, έχουν τον ελεκτικό, έχουν την... Ίσως να πάω λίγο πιο γρήγορα, α, πιο αργά εννοείται μάλιστα. Να προσπαθήσουμε λοιπόν σε χαμηλότερο επίπεδο να εξασφαλίσουμε το συντονισμό. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Φιλιππίν και ο κανονισμός του βλέπουμε ότι έχει τον όρο της διασυνο, ε, διασυνοριακής, δηλαδή διεθνικής συνεργασίας, αλλά δεν βλέπω σύνδεσμο μεταξύ του ταμείου αυτού και ταμείων ε, ή μάλλον κονδυλίων διασυνοριακών ή θεματικής συγκέντρωσης. Όταν λοιπόν λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό και το κοινωνικό ταμείο για τη διασυνοριακή συνεργασία, γιατί δημιουργούνται θέσεις εργασίας, υπάρχει μια κοινή αγορά. Πρέπει να αναπτύξουμε το μέσον ε, συνδέοντας την Ευρώπη. Πρέπει ασφαλώς σε όλα αυτά να εντάξουμε και τη θεματική συγκέντρωση. Και ας ε, αφήσω κατά μέρος το κουσουπού για να περάσω στις περιφέρειες ε, και την βελτίωση των πιστώσεων που θα πρέπει να λαμβάνουν. Οι διαπεριφερειακές ε, περιφέρειες, οι διασυνοριακές περιφέρειες θα πρέπει να έχουν αντίστοιχη χρηματοδότηση πιστεύω. Μερικές φορές έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο απασχόλησης ε, χαμηλό, ε, χαμηλή πυκνότητα πληθυσμιακή. Δηλαδή έχουν συνθήκες αντίστοιχες με τις άκρως απομακρυσμένες, απομεμακρυσμένες περιοχές. Mm. Και θα πρέπει να του δώσουμε ιδιαίτερη σημασία και προσοχή. Στρατηγικές όπως το περιβάλλον, οι μεταφορές αναπτύσσονται συχνά σε εθνικό επίπεδο. Και όταν φτάσει κανείς στα σύνορα αντιμετωπίζει δύο διαφορετικές στρατηγικές και δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει αν είναι μεταξύ τους συμβατές ή όχι. Άρα θα πρέπει να εντοπίσουμε κάποιες ε, αδυναμίες, τις όποιες αδυναμίες και να τις αντιμετωπίσουμε. Πέντε θεματικοί στόχοι είναι για μας ε, επαρκείς νομίζω ότι ίσω έξι είναι καλύτερο, αλλά το συζητούμε για τις επενδυτικές δυνατότητες και προτεραιότητες. Θα θέλαμε να ενισχυθούν, να αυξηθούν για να συμπεριλάβουν τον πολιτισμό, τις διασυνοριακές υποδομές και άλλα αντίστοιχα θέματα. Αν ε, καλυφθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ίσω δεν χρειάζεται να τα βάλουμε στο δικό μα κανονισμό, αλλά εν πάση είναι μια προσέγγιση την οποία υποστηρίζουμε. Και τελευταία σχόλια, οι κοινοί δείκτες που συμπεριλαμβάνονται θα πρέπει πιστεύω να αποτελέσουν δείκτες ως πρότυπα, που θα χρησιμοποιούνται ως πρότυπα, διότι αν τους εντάξουμε στο παράρτημα, ίσως να προ... Ε, υποθέτουν δραστηριότητες οι οποίε εξάπατος θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί για να λειτουργήσουν. Όχι, νομίζω ότι θα πρέπει να ορίσουμε κάποιε προτεραιότητε, κάποιου στόχους, με κάποιου δείκτες ε, που θα μας λένε τι πρέπει να κάνουμε μια ενδεικτική προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εσάς κύριε Σιγητά και την Επιτροπή Περιφερειών για τη συνεργασία. Ας περάσουμε στους ε, σκιώδης ηγητές. Η Μαρή Τερέζη είναι η πρώτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα φυσικά και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της και να την ευχαριστήσω κυρίως για το συνεργάσιμο και διαλλακτικό της πνεύμα έχουμε, είχαμε ήδη πολύ αγαστή συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία είναι σημαντικός μηχανισμός κατά πολέμηση της κρίσης και θα βελτιώσει την καθημερινότητά μας. η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι πέρα από τα σύνορα. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω την έκθεσή μου ε, και την έκθεση Πίπερ ε, για τον προπολογισμό ζητήσαμε 7% ναι. για την πολιτική συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα 3,48%. Αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με την προηγούμενη μας θέση και να ε, εξασφαλίσουμε πραγματική εδαφική συνεργασία, θα πρέπει να μείνουμε στην, ε, στο έτοιμά μας για 7%. Συμφωνώ με την εισηγήτρια σε ό,τι αφορά την τροπολογία 7 και το άρθρο 4. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των κονδυλίων. Στις δύο εκθέσεις που σας ανέφερα, ζητούσαμε κατανομή των κονδυλίων ανά πρόγραμμα συνεργασίας, για να αποφύγουμε να έχουμε χαμηλή απόσβεση επενδύσεων. Και σήμερα στις ε, μεθοριακές ζώνες έχουμε πολύ θετικά προγράμματα που έχουν ε, μπλοκαριστεί επειδή η ισπανική πλευρά έχει εξαντλήσει τις πιστώσεις. Γιατί δεν βρω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατανομή ένα πρόγραμμα. Έθεσα την ερώτηση, αλλά η απάντηση δεν ήταν πολύ σαφή. Το άρθρο 4 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία προβλέπει ότι η κατανομή γίνεται ένα κράτο μέλο ετησίω με βάση το δημογραφικό κριτήριο. Θα πρέπει να επιμείνουμε στο γεγονό ότι η νομιμότητα, η νομιμοποίηση μία, ενός προγράμματος είναι ε, η ωφέλεια του προγράμματος και όχι ε, το όφελο του κάθε κράτου μέλου. Το άρθρο 4 προβλέπει του τρόπου κατανομή των πιστώσεων ώστε να γίνει αυτή η κατανομή των κονδυλίων αναπρόγραμμα. Επίσης, ό,τι αφορά την ε, γεωγραφική ελαστικότητα κάποιων παρεμβάσεων εκτός του προγράμματος, είναι πολύ ανελαστική. Αν θέλουμε να κρατήσουμε το όριο των 150 χιλιόμετρων, θα πρέπει να προβληματιστούμε ως προς την αναγκαία ελαστικότητα ε, που χρειαζόμαστε για τις επενδύσεις που βρίσκονται εκτός ζώνης συνεργασίας. Ό,τι αφορά το ποσοστό συγχρηματοδότησης. Πώς ε, θα κάνουμε ελκυστικά τα κονδύλια διασυνορική συνεργασίας για ε, περιφέρειες που έχουν ε, ποσοστό ανώτερο, το 85% δηλαδή. Συνήθως έχουμε πολύ πιο περίπλοκες διατυπώσεις από τους άλλους στόχους της πολιτικής συνοχής δεν ξέρω αν τα ενάψματα που δίνουμε είναι επαρκή. Επαναλαμβάνω, χρειαζόμαστε αξιολόγηση των μέσων ε, ποσοστών ε, χρηματοδότησης για την τρέχουσα περίοδο. Γιατί με μια τέτοια αξιολόγηση θα έχουμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα για τη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά την τεχνική αρρωγή το όριο του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ είναι πολύ περιοριστικό. Είμαι υπέρ τη θεματική συγκέντρωση για να γίνει ο προγραμματισμός πιο αποτελεσματικός και να έχει πιο στρατηγικό χαρακτήρα. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα στο άρθρο 5. Και συμφωνώ με την πρόταση τη εισηγήτριας για υποβολή 5 θεματικών στόχων και όχι 4. Το παράρτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο περιλαμβάνει ένα ενδιαφέροντα κατάλογο για πιθανές δυνητικές επενδύσεις ό,τι αφορά την διαπεριφερειακή συνεργασία. Βέβαια, αν το αυτό γίνει παράρτημα του κανονισμού, θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους τρόπους συντονισμού των κονδυλίων στα πλαίσια του στόχου εδαφικής συνεργασίας. Συμφωνώ και με την προσθήκη στο άρθρο 6 της ηγετρίας για τις προτεραιότητε των επενδύσεων. Θεωρώ πάντως ότι υπάρχει ένας μεγάλο, μεγάλος απόν από τις προτάσεις αυτές. Δεν υπάρχει πολιτισμός. Θα μπορούσαμε να τροποποιήσουμε το 6 και να συμπεριλάβουμε και τον πολιτισμό στην εδαφική συνεργασία. Σε ό,τι αφορά το συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η εδαφική συνεργασία, ακριβώς λόγω της απλούς τη απλοποίηση τη μπορεί να τα χρηματοδοτήσει όλο μέσω του ΦΕΝΤΕΡ. Ήδη είναι περίπλοκοι κανόνε. Προσοχή λοιπόν να μην του περιπλέξουμε περισσότερο. Είναι σημαντικό ότι το νέο διασυνοριακό σκέλο του Κοινωνικού Ταμείου να είναι συντονισμένο με το στόχο τη εδαφική συνεργασία. Σε ό,τι αφορά του δείκτες, χρειαζόμαστε προσαρμογή του στους στόχους της εδαφικής συνεργασίας για την απλούστευση της διαχείρισης και του ελέγχου και ιδιαίτερα το θέμα ε, των ε, οργανισμών πιστοποίησης και διαχείρισης. Και εκεί χρειαζόμαστε κάποια ελαστικότητα. Η αρχή πιστοποίησης ε, μπορεί να δώσει μια εμπειρογνωμοσύνη και αρρωγή, αλλά δεν είναι σωστή η πρώτη κατάργηση, δεν ισοδυναμεί με απλοποίηση. Τέλο, τα περιφερειακά προγράμματα του ΦΕΝΤΕΡ θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα εδαφική συνεργασία και των μακροπεριφερειών. Είμαι υπέρ της αύξηση ε, των καταποκοπής ε, προκαταβολών από 15% σε 20% για το προσωπικό και συμφωνώ με την τροπολογία 20 που ζητά καλύτερο συντονισμό τη Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασίας στα επιχειρησιακά προγράμματα με τα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Πολιτικής γειτονία. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω την εισηγητρία για την αξιόλογη της έκθεση και χαίρομαι για τη σύμπνοια που υπάρχει μεταξύ μας. Σας ευχαριστώ. Φραντσέσκο Δε Άντζελης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστήσεις την εισηγήτρια, Μάνε, για όλους αυτούς τους μήνες δουλειά που κατέβαλε. Και οι συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών ήταν ιδιαίτερα επικοδομητικές. Ιδίως επειδή κατέγραψαν τις προτάσεις, τις συστάσεις, τις επιθυμίες μας. Με ιδιαίτερη προθυμία. Έτσι, το έγγραφο του Μαρτίου για το σχέδιο έκθεσης που έχουμε φτάσει να συζητούμε σήμερα καθορίζουν μια συνολική πορεία προς το, προς το στόχο της εδαφικής συνεργασίας. Με ιδιαίτερη έμφαση στην σαφήνεια. Περνάω τώρα στην ουσία λόγω χρόνου. Το σχέδιο που μας παρουσιάζει η συνάδελφο είναι βήμα προόδου για πολλούς λόγους. Κατά πρώτον, ε, μπορεί να άρει κάποιες από, από τα αμφιλεγόμενα σημεία του προηγούμενου κειμένου. Προβλέπει μεγαλύτερη ευελιξία για τους στόχους και εισάγει στοιχεία επιθυμητή και λογικής διαλλακτικότητα και απλούστευση. Το σχέδιο έκθεσης Δίνει λοιπόν μια όθηση στην εδαφική συνεργασία, φιλόδοξη, ενεργή. Και ιδίω με, την έκθεση, με την έκδοση των εκθέσεων Πίπερ και Σάντσα Σμιθ. Για το μέλλον της συνοχής ε, που θα καθορίσουν την εδαφική συνεργασία στην Ευρώπη. Εδώ υπάρχει μια δέσμευση πιστώσεων, 7% του συνολικού προπολογισμού, σημαντική. Κυρίω για, την, για τον πολιτικό προγραμματισμό των διαφορετικών ταμείων. Τρίτο σημείο, η προσέγγιση μπορεί να μας βρει σύμφωνος γιατί ακολουθεί τη γενικότερη πορεία του Κοινοβουλίου των τελευταίων ετών. Και με την έκθεση Μπάρκ είχαμε την ευκαιρία να προτείνουμε εδαφική συνεργασία με περισσότερε φιλοδοξίε, με μεγαλύτερη όθηση και από την άποψη των πόρων και του κριτηρίου τη ευελιξία, αλλά και των πολιτικών στόχων τη. Υπάρχουν βεβαίω κάποιοι ενδιασμοί και κάποιε επιφυλάξει, όμω πρόκειται για σημεία όπου πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συνεννόηση με την ε, εισηγητρία επειδή έχουμε διασφαλίσει κάποια από τα κριτήρια ευελιξία, όπω έλεγα, είμαστε ικανοποιημένοι. Όμω έχουμε πολλαπλασιασμό των εξαιρέσεων και παρεκκλήσεων που δεν εξυπηρετούν το γενικότερο στόχο τη εδαφική συνεργασία. Όπω το παρελθόν μπορεί να δημιουργηθεί ένα αποθεματικό για περιοχέ παραμεθόριε και τι εξοχώ απομακρυσμένε. Επίση, στα πλαίσια τη Στατική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 θα πρέπει να θέσουμε κάποιου Βασικού στρατηγικού στόχου, ακόμη και για την εδαφική συνεργασία. Όχι κάτι περισσότερο, αλλά και κάτι λιγότερο από ότι προβλέπεται με τους υπόλοιπους στόχους της πολιτικής συνοχής. Δεύτερο σημείο, για την πρόταση διεύρυνσης των ε, διασυνοριακών προγραμμάτων εταιρικής σχέσης καλό θα είναι να εμβαθύνουμε λίγο. Εγώ δεν έχω καταλάβει πολύ καλά τι ωφέλη θα προκύψουν στην επιδίωξη του συνολικού μας στόχου. Πέρα από το να εξυπηρετηθούν οι ενδιαφερόμενες ε, περιοχές που βρίσκονται κοντά στα σύνορα. Θα πρέπει να υπάρξει ένας, ε, μια μεγάλη προσπάθεια για τέτοιου είδους διασυνοριακή συνεργασία που όμως σε εθνικό επίπεδο μπορεί να προσφέρει μόνο μερικά ψίχουλα και όχι κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για την εδαφική συνεργασία που επιδιώκουμε. Μάλιστα έτσι η εδαφική συνεργασία θα γίνει αποκλειστικό προνόμιο κάποιων κρατών με κοινά σύνορα. Νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή η Ευρώπη να υιοθετήσει μια ενιαία προσέγγιση για τη στρατηγική των μακροπεριφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σε ένα σκηνικό που διαρκώς εξελίσσεται. Η εδαφική συνεργασία θα πρέπει να ακολουθεί τους στόχους ανάπτυξης των δύο μεγάλων ευρωπαϊκών μακροπεριφερειών. Όμως, αυτό μπορεί να μην καλύπτει τις επιμέρους ανάγκες, τις ιδιαίτερες ανάγκες των περιφερειών. Βεβαίω η συνεργασία μπορεί να είναι η μόνη κατάλληλη πηγή χρηματοδότηση, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και οριζόντια πρόθεση αυτή τη προτεραιότητα. Αυτά είναι τα βασικά σημεία τα οποία ήθελα να θίξω. Συνολικά νομίζω ότι το έργο αυτό είναι, το έργο της Ισχύτριας είναι εξαιρετικό και με αυτά τα τελευταία σημεία εφόσον κάπως αφενήσουμε, νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία με την εισηγήτρια. Πολύ καλή δουλειά λοιπόν. Με στόχους και φιλόδοξους, αλλά και πάρα πολύ σαφείς. Ευχαριστώ. Ja, danke für die Bemerkung. Der ναι, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αλφόνζη είναι η επόμενη, παρακαλώ. Ο κύριος Merci, Président. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για μας η γραφική συνεργασία συνιστά θεμελιώδη άξονα συνεργασίας και στρατηγικής για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί κοίτασμα οικονομικής ανάπτυξης. Εμείς πιστεύουμε ότι στη μονιμότητα, στους μηχανισμούς, στην ε, αδράνεια που γεννά το διασυνοριακό φαινόμενο υποκρύπτονται πολλές δαπάνες, διασπάθηση χρήματος, χαμένα λεφτά και επίσης μπορούν να αποτελέσουν παράγοντα ανάπτυξης περιφέρειας των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης σε φιλοσοφικό έτερο επίπεδο θα έλεγα ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την πολιτική αυτή που προσφέρει ε, προσθέμενη αξία ευρωπαϊκή και μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της παρουσίας Ευρώπης γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν συμφωνούμε με τον συγχυτή και την θέση της επανεκτίμησης της φιλοδοξίας μας για, τις, τη διασυνοριακή, διαπεριφερειακή συνεργασία, το 7% που έχει σημαντικά μειώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις προτάσεις της και που στις ε, προτάσεις Επιτροπής διαπιστώνουμε ότι δεν ε, ευθυγραμμίζονται με την σημασία που αποδίδουμε εμείς στην ε, υπόθεση αυτή. Τα θαλάσσια σύνορα, τα 257 χιλιόμετρα που επιβάλλει η νομοθεσία και που δεν θα πρέπει να ισχύουν για τα θαλάσσια σύνορα σε νησιωτικές περιοχές, γιατί μπορεί να ισχύσει γενικά στα θαλάσσια σύνορα, αλλά οι περιοχές οι οποίες πλήττονται κυρίως είναι αυτές που έχουν μόνο θαλάσσια σύνορα, δηλαδή τα νησιά. Και άρα, ε, αναγκαστικά και έστω και μόνο κατά εφαρμογή του άρθρου 74 της συνθήκης θα έπρεπε να εξετάσουμε μια εξαίρεση των νησιωτικών ε, εδαφών, των νησιωτικών περιοχών, ώστε να ενσωματωθούν και αυτές πλήρωσε μια πολιτική εδαφική συνοχή και συνεργασία, γιατί το αόριο αυτό που να το υπενθυμίζω, θα απέκλειε κάθε δυνατότητα συνεργασία μεταξύ τη Κορσική και των Βαλεαρίδων, γιατί μεταξύ του ε, παρεμβαίνουν μόνο 20 χιλιόμετρα, 220 χιλιόμετρα. Άρα θα μπορούσε να αναπτυχθεί αυτή η συνεργασία, ενώ θα έπρεπε να την προωθήσουμε όπω και την χερσαία περιφερειακή συνεργασία. Επίσης πολύ σημαντικό και επιφύλαξη για κατάθεση τροπολογίας όταν μιλούμε για υποδομές μεταφορών Φερρυπίν, βεβαίως οι επενδύσεις σε τοπικό επίπεδο επιτρέπουν να βελτιώσουμε σημαντικά τις ε, διασυνοριακές σχέσεις, αλλά άμεσα στην λογική αυτή ενσωματώσουμε και πολύ ε, επαχθείς επενδύσεις ε, ίσως δεν αποδώσουν όπως θα έπρεπε. Ίσως λοιπόν θα ήταν καλό να μιλούμε για επενδύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τοπικού χαρακτήρα για να μην εμπλακούμε σε προγράμματα που θα είχαν άλλες διαστάσεις και άλλη επιλεξιμότητα. Και επίσης θα ήθελα για να προχωρήσω να πω ότι η βελτίωση της ευελιξίας είναι όντως για μας μια σωστή ε, ένας επαναπροσδιορισμός, ε, δεδομένου ότι είναι πολύ ποικίλη η εικόνα παρουσιάζουν οι περιφέρειες για λόγους γεωγραφικούς καταρχάς, ορεινή, νησιωτική, παροθαλάσσια, παρόχθια, για λόγους ιστορικούς αλλά και για λόγους οικονομικούς. Η ευελιξία δεν μπορεί παρά να βελτιώσει την ε, εμφάνιση των προγραμμάτων που θα αναπτύγονται στην κάθε περιοχή. Η μακροπεριφέρεια επίσης, θα ήθελα να επισημάνω, ότι επιτρέπει τη βελτίωση του προσδιορισμού της συνεργασίας και των στρατηγικών, των μακροπεριφερειακών αυτών στρατηγικών, που μπορεί σε διάφορες περιοχές και χώρους της Ευρώπης να βρουν εφαρμογή με σημαντική ε, απήχηση στην εδαφική συνεργασία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ ιδιαίτερο στην αγαστή συνεργασία που έχουμε με την εισηγήτρια κατά την σύνταξη της έκθεσης και πιστεύω ότι υλοποίησαμε τους βασικούς μας στόχους που είναι η διευκόλυνση των, των συμπολιτών μας μέσω καλύτερης πρόσβασης σε όλες τις βασικές υπηρεσίες. Αναφερθήκατε στη σημασία που έχουν οι υποδομές και τα σχέδια υποδομών για τη διασυνοριακή συνεργασία και την εδαφική συνεργασία. Επίσης, ε, είναι ένα μέσο για την ε, συνεργασία σε διάφορα αναπτυξιακά προγράμματα μεταξύ των διαφόρων περιφερειών. Χρειαζόμαστε όμως συντονισμό πρώτα απ' όλα. Έχω ένα πρόβλημα με το άρθρο 25 του κανονισμού. Η Επιτροπή θεωρεί ότι ο βασικός εταίρος θα πρέπει να είναι και εγγυητής όλων των πληρωμών και των υπόλοιπων χωρομελών. Αυτό είναι υπερβολικό όμως και δημιουργεί τεράστιο άχθος για το βασικό εταίρο. Επίσης, δεν θα πρέπει να διευρύνουμε το πεδίο εφαρμογή των ταμείων γιατί ήδη έχει προτείνει αύξηση των κονδύλων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν χρειάζεται περισσότερη. Και τέλος, για τη μακροπεριφερειακή στρατηγική. Πιστεύω ότι χρησιμοποιούμε τη στρατηγική αυτή των μακροπεριφερειών και σε άλλα προγράμματα. Δεν χρειάζεται λοιπόν να τα αναφέρουμε και στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο συγκεκριμένο κανονισμό αρκεί να αναφέρεται η μακροπεριφερειακή στρατηγική στο γενικό κανονισμό. Ευχαριστώ. Τέσσερι ομιλητέ έχουμε ακόμη, αγαπητοί συνάδελφοι, αλλά παρακαλώ δύο λεπτά ο καθένα. Δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Ο κύριο Μάρκου Πίπερ, παρακαλώ, δώστε το καλό παράδειγμα, κύριε Πίπερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Διασυνοριακές περιφέρειες και υποδομές. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστώ την εισηγήτρια αλλά και τους κοιόδης εισηγητές ε, που έκαναν μια πάρα πολύ καλή δουλειά από κοινού. Και εν προκειμένου για, την, ε, για τον κύριο Λάζακ και την ε, πολιτική του ομάδα ECR Θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στο Connecting Europe Facility, το μέσο για, ε, συνδέοντας την Ευρώπη, στις ε, υπερσυνοριακές ε, περιφέρειες, έτσι ώστε να διατηρηθούν τα κονδύλια που έχουμε διαθέσιμα. Θα μπορούσε αυτό μέσο, δηλαδή το Connecting Europe, να ε, συνδεθεί με υπερσυνοριακές προτάσεις και να, να αναγνωριστούν προς τα αρμοδιότητες της περιφέρειας. Ναι, αυτό από πλευρά μα ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να αποτελέσει μια καλή ιδέα δει του Συμβουλίου ενδεχομένω. Ίσως ε, με την κυρία Μένερ, άλλους αρμοδίους θα έπρεπε να το συζητήσουμε αυτό. Μπορούμε έτσι να επιλύσουμε την ε, σύγκρουση. Ευχαριστώ κύριο Σόλμπρεχτ. Ευχαριστώ. Θα πρότεινα να επανέλθουμε στο 85% χρηματοδότηση. Ε, αναφέρεται στο γενικό κανονισμό, όπως είπε και ο εισηγητής από την Επιτροπή Περιφερειών. Τώρα για το διασυνοριακό χαρακτήρα στις μακροπεριφέρειες έχω σοβαρές αμφιβολίες, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το αναπτύξουμε δυστυχώς. Είναι κάπως σαφές αυτό το σημείο. Και το τρίτο, δεν αναφέρεται στο νομικό κείμενο, αλλά στο πρώτο τμήμα του κειμένου. Θα πρέπει να ληφθεί άμεσα, άμεσα απόφαση ε, για, για τα προγράμματα Urban Interact τα υπάρχοντα προγράμματα, γιατί οι άνθρωποι απασχολούνται εκεί. Θα πρέπει να ξέρουν αν στο μέλλον θα έχουν δουλειά ή όχι. Και αυτό θα πρέπει πάρα αυτά να ε, διαθετηθεί. Θα το ε, αντιμετωπίσουμε ως ανοιχτό διαγωνισμό ή ως ε, σταθερό στοιχείο. Ευχαριστώ, ο κύριος Νίλσεν. Θα είμαι και εγώ λακωνικός. Και οι Ρίκα Μάνερ και οι σκιοδησηγητές επιτελούν πολύ αξιόλογο έργο και νομίζω ότι καλό θα ήταν να διαβάσετε προσεκτικά και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών, γιατί και αυτή περιέχει πολύ εύστοχες προτάσεις. Ένα πρόβλημα που επισήμαναν πολλοί συνάδελφοι αναφέρεται στον προγραμματισμό των ε, διασυνοριακών υποδομών. Στη Βόρεια Φιλανδία, Νορβηγία και Σουηδία έχουμε συνεργασία μεταξύ ε, των περιφερειών που είναι σχετικά αεροκατοικημένε. Είχαμε στενή συνεργασία για χρόνια ολόκληρα και είχαμε πολλά προβλήματα να πείσουμε τις κυβερνήσεις μας να καταρτήσουν κοινά σχέδια, όχι μεμονωμένα εθνικά σχέδια, αλλά κοινά σχέδια μεταξύ των τριών χωρών, Νορβηγία, Σουηδία και Φιλανδία. Και πολλά σχέδια και προγράμματα που τα διαχειρίζονταν οι περιφέρειες είχαν προτάσεις ε, για, τις, ε, για, τις, ε, για τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι χώρες προκειμένου να συντάξουν, να καταρτήσουν τέτοια κοινά σχέδια. Ας μην ξεχνούμε λοιπόν και τέτοια σχέδια και προγράμματα που θα μας βοηθήσουν να πιέσουμε τις κυβερνήσεις να συνεργάζονται μεταξύ τους. Ευχαριστώ, Λάμπερτ για ολόκληρη την ομάδα. Αυτό που θέλαμε να περάσει ήταν η ιδέα τη διασυνοριακή συνεργασία ω προ την εδαφική συνεργασία. Εγώ θεωρώ ότι είναι προ τη σωστή κατεύθυνση αυτό. Όμω, στο άρθρο 19, στην τροπολογία συγκεκριμένα 19, όπου λαμβάνεται υπόψη τη διαπεριφερειακή συνεργασία και τη δυνατότητα να λαμβάνεται υπόψη και η καινοτομία και η έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα σκέφτεται να καταργήσει τις περιφέρειες έρευνας που ήταν ένα ξεχωριστό πρόγραμμα. Θα πρέπει κάθε περιοχή να γνωρίζει την εξειδίκευσή της, να την ορίζει και να αναζητά εταίρους Έτσι μπορεί να καθορίσει την ποιότητά της, στατιστικώς από τα αποτελέσματα το πώς θα χρηματοδοτηθεί για να κατέχει μια θέση στην Ευρώπη. Όμως το πρόγραμμα αυτό δεν υπάρχει πλέον στην πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Θα πρέπει όμως να προωθήσουμε την διαπεριφερειακή συνεργασία. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα ευρύτερο. Μπορούμε να διευκολύνουμε τα πράγματα από τη μια. Και από την άλλη, για την επιχειρησιακή συνεργασία, θα πρέπει να πάρουμε κάποια τμήματα από, το, από άλλα κομμάτια του Ταμείου. Ε, Πάντω θα πρέπει κάτι να κάνουμε εδώ για, τις, ε, για την περίπτωση τη έρευνα, αυτή την παράγραφο και όχι αλλού, για να μην λέμε εκ των υστέρων συγγνώμη. Ε, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επειδή είναι μεγάλη χρονική πίεση, έχουμε κάποια σχόλια. Αλλά θα δώσουμε απευθεία το λόγο στην συγκήτρια. Σα ευχαριστώ, κυρία Μάνερ. Θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, πολύ γρήγορα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για τα σχόλιά τους, ιδιαίτερα χρήσιμα και επικοδομητικά. Και Θα συζητήσω με τον κύριο Πίπερ, τον κύριο Όλμπριχτ και να τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή, γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάντως ιδιαιτέρως και όλα τα σχόλια θα τα λάβω υπόψη μόλις υποβάλουμε τις νέες τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μέχρι την 31η Μαΐου 6 το απόγευμα ε, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Περνάμε στο σημείο 8 Μαρία Ριγκόγεν Πέρε, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Έχετε το λόγο. Muchas gracias, muchas gracias, Presidenta, viendo lo, lo avanzado de esta hora y con... Ευχαριστώ. Ε, δεδομένου του προχωρημένου της ώρας ε, και μετά από μια πολύ έντονη συζήτηση και πολύ ε, συγκινησιακά φορτισμένη από το πρωί, θα προσπαθήσω για να κατευνάσω τα πνεύματα, να περάσουμε σε ένα θέμα της 31 μία τροπολογίες που έχω υποβάλει σε ένα έγγραφο. Είναι ο καρπός πολύ καρποφόρος συζητήσεων που είχαμε στην Επιτροπή και ανταλλαγή απόψεων με τους και οδησηγητές. Θα ήθελα να περάσω κατευθείαν στο σχολιασμό των νέων τροπολογιών για να επιταχύνουμε και να διευκολύνουμε και τη συζήτηση. έχω προτείνει κάποιες αλλαγές επιμένοντας τις προτεραιότητες. Μία προτεραιότητα είναι η προώθηση της ε, ενεργούς και διαρκούς ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, προλάβουμε και να προβλέψουμε την προσαρμογή των εργαζομένων στην αγορά εργασίας. Και φυσικά να προσέξουμε ιδιαίτερα τις ε, επιχειρήσεις που έχουν ε, επιχειρήσεις, ε, τις περιφέρειες που έχουν επιχειρήσει αναδιάρθρωση ή ε, που βιώνουν τη μετεκατάσταση των επιχειρήσεων. Θέλουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των εργαζομένων χάρη στην διασυνορική ολοκλήρωση των αγορών εργασίας. Επίσης, επισημαίνουμε την ανάγκη κατάλληλης παρέμβασης ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων κοινοτήτων σε ό,τι αφορά την παιδεία, τη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων και την κατάρτιση. Η κοινωνική ένταξη είναι ένα άλλο σημαντικό σημείο ε, και η ένταξη των ε, μεταναστών. Ένα στόχος που είχε εξαφανιστεί από τη νέα πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά περιλαμβανόταν στην προηγούμενη πρόταση του 2006. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι προσπάθησα να πηχήσω τις ανησυχίες ε, πολλών σχεδόν εισηγητών και να αναφέρω την ανάγκη συμπληρωματικότητας των ταμείων. Αηφόρος ανάπτυξη των πόλων, για παράδειγμα, πρότεινα το ποσοστό 5% να αφιερώνεται στο θέμα αυτό. Επίσης, θέλουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να στηρίξει την αηφόρο ανάπτυξη της πόλη. Θα καταθέσω ακόμη λίγες τροπολογίες τις επόμενες μέρες για τη χρήση των μικροπιστώσεων, για παράδειγμα, μεταξύ των πιθανών χρηματοπιστωτικών μηχανισμών, για τη χρηματοδότηση μέτρων και πολιτικών. Θα ήθελα να αναφέρω τις ε, περισσότερο ανεπτυγμένες περιοχές, τον κατάλογο θεμάτων για διασυνοριακή συνεργασία, την συνέπεια και συμπληρωματικότητα μεταξύ των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και των δράσεων της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης για την Αλλαγή και τις ε, βασικές παρεμβάσεις. Επίσης θα υποβάλω μια τροπολογία και για τους δείκτες. Αυτά Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ελπίζω να ήμουν αρκετά σύντομη, ώστε να προλάβουν και οι υπόλοιποι συγγετές που έχουν σημειώσει στην ημερήσια διάταξη να μας τα παρουσιάσουν. Ευχαριστώ. Ε, Από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγητριά μας για την ε, καταπληκτική προετοιμασία που έκανε ε, για την έκθεσή της και για την ε, πολύ εργαστή συνεργασία. Πολλές παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις που υποβάλαμε στις συναντήσει με την εισηγήτρια ελήφθησαν υπόψη τελικά στην έκθεσή της και την ευχαριστώ ιδιαίτερος γι' αυτό. Είμαι πολύ ικανοποιημένη γιατί σε πολλά σημεία η εισηγήτρια αναφέρθηκε ε, στους νέους, στις γυναίκες, στους ηλικιωμένους, στην ιδιαίτερη κατάστασή τους στην αγορά εργασίας. Χαίρομαι που γίνεται μία και αυτό του θέματος. Επίσης αναφέρθηκε η ανάγκη να βοηθηθούν οι νέοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας αμέσως μετά την αποφύτισή τους. Άλλο σημαντικό θέμα για μένα είναι ε, και για όλες τις γυναίκες φαντάζομαι το θέμα της ε, άνευ προβλήματος ε, επαναφοράς στην αγορά εργασίας μετά την άδεια μητρότητας. Σημαντικό που αναφέρεται. Επίσης το θέμα της, ε, των μισθολογικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι πολύ σημαντικό. Ένα άλλο κέριο ζήτημα είναι κάτι που συμπεριέλαβε στις τροπολογίες και αφορά τη διεύρυνση των επενδυτικών προτεραιοτήτων από 4 ε, σε 6. Γιατί πολλές φορές οι περιφέρειες ζητούν περισσότερη ελαστικότητα και επίσης ε, περιορίζεται σε 10% η συμμετοχή κάθε κατηγορίας περιφερειών. Νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει και θα ικανοποιήσει τους δικαιούχους. Θέλουμε αυτά τα κονδύλια να αξιοποιηθούν και πραγματικά να έχουν κάποιο αποτέλεσμα για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, για την καταπολέμηση της φτώχειας, για τη βελτίωση της απασχόλησης και ούτω καθεξής. Είναι πολύ σημαντικό να αναφέρονται τα θέματα της καταπολέμησης της φτώχειας, τα προβλήματα της απασχόλησης, οι κοινωνικές διαφορές. Στη διάρκεια της συζήτησης και σε συναντήσεις που είχαμε με εκπροσώπους των περιφερειών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, με δικαιούχους, ακούσαμε κάποιες ανησυχίες που έχουν και αφιβολίες ό,τι αφορά την ελάχιστη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική εκταμίευση. Ε, νομίζω ότι φοβάμαι μήπως η βελτίωση αυτή του ελάχιστου ποσοστού οδηγήσει σε περιορισμό των ποδηλίων για κάποιες ε, επενδύσεις στις υποδομές, στις βασικές υποδομές, όχι μόνο τους αυτοκινητοδρόμους, γενικές υποδομές ε, που βοηθούν και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην καλύτερη θέση των επιχειρήσεων. Ας το προσέξουμε λοιπόν αυτό. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι να αναφερθεί η βοήθεια προς τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, γιατί αυτές οι επιχειρήσεις είναι που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Οπότε μια στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για τις επιχειρήσεις αυτές, όχι μόνο για την κατάρτιση, αλλά γενικότερα για τις επιχειρήσεις, είναι πολύ σημαντική. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι μόλις σήμερα, τουλάχιστον στο δικό μου γραφείο, μόλις σήμερα ε, έλαβα την γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών παρόλο που την είχαμε ζητήσει επίμονα. Γιατί και η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειών περιλαμβάνει παρατηρήσεις και προτάσεις για τροπολογίες που φαντάζομαι στη συνέχεια θα ληφθούν υπόψη. Πάντως α, χαίρομαι και νομίζω ότι όλοι ενδιαφερόμαστε να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των στόχων, γιατί αυτό περιμένουν από εμά οι συμπολίτε μα. Περισσότερε θέσει εργασία, ποιοτικέ θέσει εργασία, οι νέοι που ονειρεύονται να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα προσόντα και τα εφόδια που συγκέντρωσαν στη διάρκεια των σπουδών τους και να μπορέσουν να τα χρησιμοποιήσουν σε μια θέση απασχόλησης. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο για όλους. Να έχει αποτελέσματα το έργο μας και να δημιουργήσει τα θεμέλια για τη βελτίωση της κατάστασης. Γι' αυτό θέλουμε μια έκθεση που θα είναι καλή, γιατί αυτό περιμένουν πραγματικά όλοι. Ευχαριστώ θερμά την εισηγητρία. Η Ραμόνα Μανέσκο απο... απουσιάζει, ο λόγος στην κυρία Σρέτερ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Όντως ε, έχει συμπεριλάβει μια σειρά από τις προτάσεις μας. Την ευχαριστούμε θερμά. Πρόκειται για σημεία στα οποία πιστεύω θα μπορούσαμε ε, να καταλήξουμε σε μια κοινή διατύπωση κυρίως για το 5% που θεωρώ πολύ σημαντικό στο άρθρο 6, ωστόσο νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσαρμογή. Η μικροχρηματοδότηση, ναι, καλό είναι που ενσωματώθηκε το άρθρο 43 είναι αυτό το οποίο δεν με ικανοποιεί τόσο γιατί προσπαθείτε να κάνετε πιο ευέλικτες διαδικασίες, αλλά δεν νομίζω ότι τα έχετε καταφέρει τόσο καλά. Η ευελιξία αυτή που προτείνεται ασφαλώς θα ικανοποιεί μάλλον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτό το σύστημα της συγκέντρωσης. Πρέπει με τις έξι προτεραιότητες, εφόσον ή ιδάλλως μία-δύο, να προχωρήσουμε κατά τρόπο ευέλικτο με τα προγράμματα. Επίσης, ε, είναι σωστό ότι πρέπει να ενσωματωθεί και το θέμα της ε, αποδημίας, της εγκατάλειψης των περιφερειών στο κείμενο. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ να σας ότι ξέρετε πολύ καλά το θέμα σας, αλλά το έχουμε συζητήσει και πολύ καιρό τώρα. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόταση. Μπορεί κανείς να επισημάνει ποια είναι τα θετικά σημεία, διαφοροποίηση διαφόρων ομάδων ε, πολιτών, νεολαία, φερρυπίν, που υποστηρίζουμε ιδιαίτερως, μετανάστες βεβαίως. Πολύ σημαντικό. Θα ήταν ε, μάλιστα κακό να έχουμε λησμονήσει αυτές τις διαφοροποίησεις σε ομάδες. Ε, βλέπουμε ότι η έκθεση εξετάσει τα θέματα από κάτω προς τα άνω και αυτό είναι θετικό, επί παραδείγμα το θέμα των μικροπιστώσεων για τις συγκεντρώσεις. Δεν είναι τόσο θερμή υποστηρίκτια των ε, ποσοστών όποια και είναι αυτά. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να περιοριστούμε σε κάποια ποσοστά ή καλύτερα να επαληθεύσουμε αν υπάρχει δυνατότητα για μια διαφορετική μεταβλητή, αν δεν τα μειώσουμε. Για τα αστικά κέντρα. Θα ήθελα να πω ότι όλοι οι συγκητές που είχαν μέχρι τώρα να ασχοληθούν με το θέμα αυτό θα ήταν καλό να καθίσουν μαζί και να κάνουν προτάσεις συμβατές μεταξύ τους για το πώς χειριζόμαστε το θέμα των αστικών κέντρων. Και είναι βεβαίως κατανοητό ότι υπάρχουν διαφορετικά κομμάτια που αφορούν τα αστικά κέντρα στην κάθε έκθεση, αλλά να είναι τουλάχιστον μεταξύ τους συμβατά, να μην έχουμε ασυνέπεια στην τοποθέτησή μας. Θα ήταν κακό αυτό. Άρα θα πρέπει να γίνει και σχετική προσαρμογή στα συμπεράσματα των επιμέρους εκθέσεων. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Φανίστελ Ρούι. Πολύ σύντομα δύο σχόλια. Ξέρω ότι επαναλαμβάνω αυτά που είπα και νωρίτερα. Πρώτα απ' όλα, μήπως μπορούμε να διατυπώσουμε την επιθυμία για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση Ταμείου Συνοχής, Ταμείου Κοινωνικού Ταμείου, Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης ως μέσον. Ε, μια ολοκληρωμένη λοιπόν προσέγγιση. Γιατί βλέπουμε ότι δεν κολλάει. Άλλη είναι η οπτική γωνία, άλλε είναι οι προθέσει, η επικοινωνιακή τοποθέτηση. Και αν μιλήσω, Φερρυπίν, με κάποιον ειδικό για τα γερμανικά κρατήδια, τα Λέντερ, κάποιον που ασχολείται με τα θέματα τη περιφερειακή ανάπτυξη ή που ασχολείται με το κοινωνικό ταμείο ή με το ταμείο συνοχή. Ο κάθε ένα από αυτού δεν γνωρίζει του άλλου, δεν ξέρει ποιο ασχολείται με τον άλλο τομέα. Κάνουν, διαφορετικά, κάνουν τα ίδια πράγματα αλλά χωριστά. Εγώ θα ήθελα όλοι αυτοί να κάνουν τη δουλειά από κοινού. Αυτό είναι ο στόχο τον οποίο τίνω, δηλαδή να έχουμε να κάνουμε με ένα χώρο που θα λαμβάνει αυτές τις ε, αποφάσεις και θα προωθεί τα θέματα αυτά. Γιατί ωραία είναι αυτά που λέμε, αλλά δεν έχουμε κοιτάξει πώ μπορούμε να τα ευθυγραμμίσουμε. Μιλάμε για πολλά πράγματα, μιλούμε για το κοινωνικό τμήμα κτλ. Ε, τα συζητάμε, συζητάμε για το κουπουσού και μετά τα αφήνουμε. Πρέπει να τα συζητήσουμε, πρέπει να τα μελετήσουμε, πρέπει να καταθέσουμε τροπολογίε. Και επίση για την ε, ευελιξία, είπε και ο Γιάννα. Γιατί δεν και καλά να ε, κολλάμε σε αυτό το 52% ας δείξουμε, ας ενσωματώσουμε και μια μέθοδο ευελιξίας, ας τα αφήσουμε πιο ελεύθερο. Και στη τελευταία ανάλυση, αν ένα κράτο μέλο αναλαμβάνει την ευθύνη ε, τη δική του πολιτική, τη δική του επιλογή προ τη μία την άλλη κατεύθυνση, και στο Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ανάπτυξη Υπαίθρου και στο Κοινωνικό Ταμείο, όλα αυτά πρέπει να, ε, πρέπει να αφήσουμε να λειτουργήσουν φυσιολογικός πόσας, μην τα διαλύουμε εμείς. Μην ξεχνάμε ότι εμείς έχουμε γνωμοδότηση μόνο για την Επιτροπή Απασχόλησης, άρα θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις δικές τους ε, κατευθύνσεις και επιλογές περισσότερο. Η συγκήτρια βεβαίως έχει τον πρωταρχικό ρόλο σε αυτό, οι συντάκτες και οι συγκήτριες, αλλά ε, ας, ρίξουμε και, ας κοιτάξουμε το θέμα και από αυτήν την άποψη. Καλώς λέει η Πρόεδρος, άρα θα το συζητήσετε μεταξύ σας. Η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την έκθεση, για την έκθεσή της. Να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία που δεν έχουν γίνει αντιληπτά. Τροπολογίες 9 ε, και 11 για ορισμένες από τις επενδυτικέ προτεραιότητες. Μην ξεχνάτε ότι οι επενδυτικέ προτεραιότητες είναι στόχοι προ υλοποίηση και δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ε, δράσεις που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τις ε, διαχειριστικέ αρχέ. Αυτό είναι μια αρχή που ισχύει για όλα τα ταμεία. Τροπολογίες 12 και 13 ίσως παρά είναι περιοριστικά τα θέματα. Αναφέρονται η Ρωμά. Δίνεται έμφαση σε κοινωνική ένταξη και ένταξη στην απασχόληση, ενώ οι εμπειρογνώμονες συμφωνούν ότι η ένταξη των Ρωμά θα πρέπει να αναφέρει και άλλες υπηρεσίες, υγεία κτλ. Να μην περιοριστούμε μόνο στην κοινωνική ένταξη και στην απασχόληση, γιατί ίσως υπερ, περιορίσουμε υπερβολικά α, τις επενδύσεις το θέμα της ένταξης είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να διατηρηθεί. Θεματική συγκέντρωση, ελαστικότητα και φιλοδοξία. Θέλουμε τα κονδύλια να τα εστιάσουμε σε μικρότερο αριθμό. Θα αυξήσουμε την απήχησή τους, την, ε, τον αντίκτυπο που θα έχουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό είναι και το ζητούμενο. Σε ό,τι αφορά το 5% που προσθέθηκε για την τοπική ανάπτυξη. Φαίνεται ότι υπάρχει μια διαφορά τώρα μεταξύ του ΦΕΝΤΕΡ και του ΕΚΤ. Θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι συνεπείς μεταξύ τους οι διάφορες διατάξεις, να μην υπάρχουν αντιφάσεις. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 28, εκεί η συγγήτρια προβλέπει ιδιαίτερο οριζόντια αποστολή για το ΕΚΤ Νομίζω ότι έχει νόημα να είναι οριζόντια αυτή η αποστολή και όχι μόνο να είναι αποστολή για το ΕΚΤ για ορισμένα είδη περιφερειών. Αυτό θα πρέπει να το ξαναεξετάσετε. Προς το παρόν αυτά, λόγω της πίεσης χρόνου, υπάρχουν κάποιες τεχνικές παρατηρήσεις, αλλά μπορώ διμερώς να το συζητήσω με την εισηγήτρια, αν δεν έχετε αντίρρηση. Γιατί, παραλαμβάνω, έχουμε μείνει λίγο πίσω, προτιμώ να ολοκληρώσω εδώ. Η εισηγήτρια έχει για ένα λεπτό τον καιρό να ανακεφαλαιώσει. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα σχόλια. Όντως ε, ήταν πολύ ωραίο το έργο, άκουνες οι και μεγάλη συνεργασία. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε την γνωμοδότηση για το ταμείο αυτό. Συμφωνώ με το σχόλιο του Λάμπερτ ε, ε, περί συμπληρωματικότητας των ταμείων. Αλλά μην ξεχνάτε ποια είναι η αποστολή του ΕΚΤ όσοι ασχολούνται με την πολιτική συνοχή θα πρέπει να ξέρουν το ιδιαίτερο χρέος του κάθε ταμείου, γιατί ο στόχος είναι κοινό, η κοινωνική ευημερία, η ένταξη, αλλά κάθε ταμείο έχει συγκεκριμένη αποστολή. Συμφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις τροπολογίες 11 και 12. Δεν αναφερόμαστε κατά ανάγκη στους Ρωμά όταν μιλούμε για την ένταξη. Καλώς. Ισχύει η ίδια προθεσμία και για την έκθεση αυτή, 31 Μαΐου 6 ε, το απόγευμα και περνάμε μέσα στη γνωμοδότηση ε, της ε, κυρίας Χακάεβα Χουσμένοβα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα πρέπει δυστυχώς να περικόψω σε μεγάλο βαθμό την ε, παρουσίασή μου λόγω του χρόνου. Πάντως θα προσπαθήσω να Αναφέρω τα κύρια σημεία, τα διορθωτικά ταμεία, ταμείο συνοχή περιλαμβάνοντα τα πλέον αποτελεσματικά μέσα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ανάπτυξη και θέσεων εργασία, την αύξηση τη ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία και τη στήριξη των μέσων μαζική ενημέρωση. Πιστεύω λοιπόν, ω εκ τούτου, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η χρηματοδότηση για τη συνοχή, όπω άλλωστε έχουμε ζητήσει η οικονομική, κοινωνική, εδαφική συνοχή, η επιτεύξη των στόχων του 2020 είναι πολύ σημαντική. Ωστόσο, η οικονομική κρίση έχει θέσει σε μια δυσμενή μάλλον κατάσταση της μικρομεσαίας επιχειρήσεις. Πολλές ήταν οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπόρεσαν να λάβουν χρηματοδότηση και η απουσία επαρκών πόρων δεν επιτρέπει την καινοτομία, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, την βελτίωση της παραγωγικότητας του εκ τούτου, την απασχόληση, την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Και γι' αυτό χρειάζονται κατεπήγοντα μέτρα για να βελτιωθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε πηγές χρηματοδότησης. Τα κατά μία μπορούν να προσφέρουν ε, αυτή τη χρηματοδότηση μέσω μετοχών, εγγύσεων και δανείων. πρέπει να ενισχυθεί αυτή η πρακτική με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της παραγωγικότητας, αλλά θα πρέπει να αποφεύγονται οι περίπλοκες διοικητικέ διαδικασίε και σημαντικέ διαφορέ μεταξύ των διατάξεων που εφαρμόζονται αντίστοιχα από τι διαχειριστικέ αρχέ και του ενδιάμεσου φορεί. Αυτό έχει συνέπεια την ε, χαμηλή απορρόφηση κονδυλίων και τη δυσκολία στην αξιοποίησή του. Ρωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώ μπορεί να βοηθήσει σε μια καλύτερη αξιοποίηση και αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών πολιτικών για να βελτιώσουμε την εικόνα τη ευρωπαϊκή οικονομίας, κυρίω στον χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, ωστόσο, πιστεύω ότι η δυνατότητες που προσφέρονται, τα μέσα που διατηθούνται θα πρέπει να εφαρμόζονται σε ευρύτερη βάση, να προσφέρονται σε ευρύτερη βάση τα κράτη-μέλη με στόχο την ε, αποφυγή της ε, επιφανειακής μόνο βελτίωση κατάστασης με στόχο να προωθηθεί μια ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής κατάστασης. Η νομοθεσία πρέπει να απλουστευθεί. Και αυτό σε κάθε επίπεδο για να δούμε απτά αποτελέσματα να αποφύγουμε τις περίπλοκες διαδικασίες, τις ε, ε, βραδίες διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο που επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ως γνωστόν έχουν απειρουσμένους πόρους. Και εν τέλει θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στην καλύτερη συνεργασία, τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ εθνικών και περιφερειακών ε, αλλά και ευρωπαϊκών επιπέδων με στόχο την ε, υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το 2020, ορίζοντας το 2020 έχει τεράστια σημασία για την, ε, ευρωπαϊκή οικονομία και σε αυτό μπορούμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο μικρομεσαίε επιχειρήσει. Άλλα θέματα όπω οι μεταφορέ, η ενέργεια, η ευρυζωνικότητα, η καινοτομία, η έρευνα και ανάπτυξη είναι θέματα που θα ήθελα επίση να συζητήσουμε μαζί σα και ελπίζω οι συγκητέ να βοηθήσουν ε, να βελτιωθεί το κείμενο, το σχέδιο αυτό κειμένου που πιστεύω θα οδηγήσει εν τέλει σε ένα καλό ε, πλήρε κείμενο όταν θα έχουμε ολοκληρώσει τη συζήτηση μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Βίγκλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν θα επαναλάβω τα σημεία στα οποία συμφωνώ με την συγκεκριμένη λόγω τη έλλειψη χρόνου. Έχει επισημάνει πόσο σημαντικές είναι οι μικρομεσέ επιχειρήσεις για τη δημιουργία νέων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ιδιαίτερα πρέπει να μεριμνήσουμε για αυτές. Βέβαια το ζήτημα της γραφειοκρατίας που επισημάνει είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χρειάζεται βελτίωση της προσβασιμότητας στα κονδύλια, προστασία της πνευματικής διοκτησίας και άλλα αντίστοιχα ζητήματα. Ένα δύο σημεία ήθελα να υπογραμμίσω, τα οποία θεωρώ σημαντικά. Είναι πολύ σημαντικό να Ε, αναφερθούμε σε καλούς ορισμούς, σε σωστούς ορισμούς το δυναμικό ανάπτυξης θα ήταν επικίνδυνο να περιγραφεί κατά τρόπο που θα απέκλεινε από ότι ο βασικό ορισμό είναι μεγάλος ο κίνδυνος λοιπόν ε, γιατί 99% των επιχειρήσεων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτονται από αυτή την έννοια όλες οι επιχειρήσεις ουσιαστικά και ως εκ τούτου εάν διευρυνθεί ο ορισμός τόσο να καλύπτει όλες τις επιχειρήσεις δεν θα έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια διαφοροποίηση μεταξύ του ποιο μπορεί να υποφεληθεί από τα προγράμματα και σε αυτό πρέπει ιδιαίτερα να φροντίσουμε να έχουμε σαφείς περιγραφές, σαφή κριτήρια. Το πρόγραμμα 2020 έχει ήδη μέτρα προβλέψει για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων το 2014. Εμεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, με την κατάλληλη πρικοδότηση στον προπολογισμό, αν και υπάρχει και περιθώριο ε, λιτότητα πιο αυστηρών διατάξεων, όπως πριν ε, στο σημείο που αναφέρεται ότι μπορεί η προτίμηση να δίνεται στο καταλληλότερο επίπεδο, το περιφερειακό επίπεδο για την υλοποίηση των ε, προγραμμάτων. Ε, Πάντω, όπω είπα, υποστηρίζω την ιδέα για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, την ιδιαίτερη υποστήριξή του, ιδιαίτερα την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δι, στην διεθνοποίηση αυτών με νέα επιχειρησιακά πρότυπα που θεωρώ βεβαίως ότι θα πρέπει να τα αντιλαμβανόμαστε στο δυνατόν πιο ευρέως, στην ευρύτερη έννοια του όρου. Η εσωτερική αγορά επίσης πρέπει να μετατραπεί σε μια εσωτερική βεβαίω αγορά, αλλά να βοηθήσει και την διεθνοποίηση, να δώσει περισσότερες δυνατότητες ε, διάθεσης προϊόντων, ε, ανάπτυξης της για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. κέντρα ενημέρωσης, πόρταλς ε, ε, γνώσεων ε, και υπηρεσίες που τι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να αποτελέσουν σημεία κέντρα υποστήριξης των προσπαθειών τους και της ανάπτυξής τους. Το ENS είναι ένα καλό μέσο, ένα καλό εργαλείο υποστήριξη και ενημέρωση δεν το έχουν αναπτύξει όλα τα κράτη-μέλη όπω θα έπρεπε. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιμείνουμε ιδιαίτερα σε αυτή τη διάσταση. Τη δικτύωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει πολύ μεγάλη σημασία και όχι μόνο για την πρόσβαση στην αγορά. Αλλά βέβαια όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με την κατάλληλη οργάνωση, Οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Ε, θα πρέπει να ενθαρρύνονται να βελτιώνονται και να αποθαρρύνονται από ασφαλμένη αξιοποίηση των προγραμμάτων, ενδεχομένως και με κυρώσεις. Όλα αυτά πάντοτε με ε, τη δικτύωση, η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τον ενδιαφερόμενο, τον πελάτη δηλαδή, και βέβαια πάντα σε καλή συνεργασία μεταξύ μα πιστεύω ότι μπορούμε να καταθέσουμε καλέ τροπολογίε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Μάνκα είναι εδώ για να μα ε, απαντήσει εκ μέρου των συλληστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Μόλκοβα, η σκέδωση ηγετρία, βρίσκεται καθοδόν προς τις Βρυξέλλες αλλά μου ανέθεσε να την αναπληρώσω. Κανονικά είναι στα σλοβακικά τα, οι σημειώσει τη σκιώδου ηγήτρια. Δεν έχουμε όμω σλοβακική σήμερα διερμηνία. Θα μιλήσω λοιπόν τσεχικά. Η σκιώδη ηγήτρια συμφωνεί με τι βασικέ ανάγκε των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ανάγκη εξασφάλιση πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Βέβαια, ενάψεις κρίσης έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες ε, παροχής δανείων και γι' αυτό έχει περιοριστεί αισθητά η πρόσβαση των επιχειρήσεων στις ε, πιστώσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια μέτρα για να ενισχύσουμε αυτή την πρόσβαση, γιατί χάρη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Η συγγήτρια πιστεύει ότι Καλό θα ήταν να μείνουμε στην οδηγία της 16 Φεβρουαρίου του 2011 σε ό,τι αφορά τις υπέρημερες πληρωμές. Δηλαδή, οι κρατικές αρχές θα πρέπει να καταβάλουν τους οφειλές τους μέσα σε 30 μέρες. Η κατάσταση όμως είναι πολύ ανησυχητική σε πολλές χώρες μέλη. Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, η κατάσταση είναι δεινή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μερικές φορές παρατείνουν μέχρι και κατά πέντε μήνες αυτή την προθεσμία και οι συνθήκες αυτές πολύ συχνά οδηγούν σε χρεοκοπία τις επιχειρήσεις αυτές Άλλο σημαντικό θέμα είναι η καλύτερη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιφερειακές αγορές. Είπαμε ότι καλό θα να δημιουργηθεί ένα δίκτυο διαπεριφερειακό που θα δίνει πληροφορίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όποια χώρα και βρίσκονται. Ευχαριστώ Γιάννα Μιράντα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σε χαρώ καταρχήν την εισηγητριά μας γιατί λόγω της κρίσης είναι πολύ σημαντικό ένα τέτοιο πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επιχειρηματικότητα σημαίνει ανάληψη κινδύνου, σημαίνει άνοιγμα, σημαίνει καινοτομία. Σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες όλη την Ευρώπη ταλανίζονται από την κρίση, ε, είναι υπερχρεωμένες και εξαιτία αυτή τη ε, υπερβολική χρέωση δεν έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα, σε χρηματοδότηση, για να μην αναφέρουμε και όλε τι ε, διοικητικέ διατυπώσει, στη γραφειοκρατία και του διοικητικού περιορισμού που αντιμετωπίζουν. Και μάλιστα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στα σύνορα ε, αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Γιατί όταν ε, μια επιχείρηση βρίσκεται στα σύνορα αντιμετωπίζει και θέλει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της και στη γειτονική χώρα, αντιμετωπίζει πολύ μεγαλύτερη γραφειοκρατία και πολύ περισσότερους διοικητικούς φραγμούς. Μιλήσατε για ανάγκη συνοχή και συμπληρωματικότητα των ταμείων και των διαφόρων κονδύλιων. Συμφωνούμε με το στόχο αυτό και φυσικά συμφωνούμε και με την ανάγκη ε, σύνταξη καταλόγου των υπαρχών προγραμμάτων και μηχανισμών για να αποφύγουμε την επικάλυψη γιατί ο γενικός στόχος είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και μάλιστα μιλούμε για θέσεις απασχόλησης για συγκεκριμένες κοινότητες, γιατί με την τεράστια ενεργεία που μαστίζει σήμερα την νεολαία θα πρέπει η βελτίωση της απασχόλησης να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους. Γιατί μερικές φορές η ενεργεία των νέων σε κάποιες χώρες μέλη φτάνει και το 50%. Ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι πολλές φορές η λύση για τους νέους αυτούς. Επίσης, να μην ξεχνούμε και την κατάσταση των μεταναστών, που όλους παραδόξως αποτελούν ε, μεγάλο τμήμα του εργατικού δυναμικού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Είναι πολύ θετικό και δυναμικό αυτό το στοιχείο των μεταναστών ε, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταπολεμήσουμε την ξενοφοβία. Μίλησε κάποιος πριν για έλλειψη υγειονομικού συστήματος. Υπάρχουν υγειονομικά συστήματα που αποκλείουν τους μετανάστες. Αυτό θα πρέπει να τα στελιτεύσουμε γιατί αν δεν επιτρέπουμε πρόσβαση στην υγεία στου μετανάστε, πώ θα έρχονται να εργάζονται στι μικρομεσαίες επιχείρησει μα. Επίση, ανάγκη χρηματοδότηση, πολύ σωστά το αναφέρετε, είναι ζωτική σημασία για να αναλάβει ένα επιχειρηματίας τον κίνδυνο να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση. Επίση, τα προγράμματα για του Νέου επιχειρηματίες και το Erasmus Mundus, που αναφέρεται από τον εισηγητή επί της ουσίας της Επιτροπής Ήτρε, τον κύριο Ρούμπιχ. Αυτά και θα συμβάλλουμε και εμείς με τροπολογίες. Ο, Βαν, ο Λάμπερτ Βανίσελ Ναι, πολύ σύντομα. Και ευχαριστώ για τις προτάσεις. Μια σχόλια. Θα γίνει συζήτηση από ό,τι φαίνεται το Στρασβούργο του, στην Ολομέλεια. Η πρόταση της Ήτρε υποστηρίζεται από διάφορες ομάδες και ιδιαίτερα η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη χρήση διαρθρωτικών ταμείων. Στρέφομαι και προς τους συναδέλφους και συντονιστές και τους ζητώ να παρακολουθήσουν το θέμα αυτό, να μείνουν μέσα στη συζήτηση ώστε να προσφέρουμε και τις μα. μας Πρώτον. Δεύτερον, ίσως είναι σημαντικό να ενσωματώσουμε και κάποιες από τις νέες μας ιδέες, νέες ιδέες που ήδη προβλέπονται στον κανονισμό στους νέους ε, κανονισμούς. Ίσως μπορούμε να είμαστε πιο επιθετικοί. Να πούμε ναι, μπορούμε να έχουμε νέα χρηματοπιστωτικά, χρηματοπιστωτικά μέσα, γιατί δίνεται η εντύπωση ότι ο καθένα μπορεί να αντλήσει κονδύλια από τα περιφερειακά ταμεία. Δεν είναι αλήθεια όμως αυτό, διότι πρέπει να προσφέρει κάποια καινοτομία αυτό που πράττει για να χρηματοδοτηθεί από τα περιφερειακά ταμεία. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι καλό να είναι ξεκάθαρα αυτά τα πράγματα. και πρόκειται για μικρομεσαίε επιχειρήσει μόνο και όχι για μεγάλου ομίλους ε, επιχειρήσεων. Εν πάση περιπτώσει, όσο είναι η διατύπωση τέτοια που να αποσκοπεί στην ε, συμπλήρωση της, της τη της ΣΥΤΡΕΑ, ίσως μπορώ και να βοηθήσω. Μάλιστα, αν κατάλαβα καλά, ο κύριος ε, Νεφανής Ρόι προτείνει την βοήθειά του, προσφέρει χείρα βοηθεία στην συντάκτρια. Δεν ξέρω αν είναι εξάντε ή εξπόστη η εξποστη αιρεσιμοτητα της βοήθειας που προσφέρετε κύριε Φανίστηλ Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε εσείς κάτι. Πρόεδρε, ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλες τις προτάσεις, ε, τις συστάσεις, τις υποδείξεις. Με επιβεβαιώνουν στην επιλογή μου, στην επιλογή κατεύθυνσης. Περιμένω συγκεκριμένε προτάσει πλέον, έτσι ώστε να βελτιώσουμε ουσιαστικά το κείμενο. Καλώ, λέει η Πρόεδρο. Έχουμε μέχρι τι 15 Μαου, τι 12 το μεσημέρι, την προθεσμία για την κατάσταση των προλογιών. Και τώρα περνάω στο τελευταίο θέμα τη ημερήσια διάταξη, που είναι η εξέταση του εγγράφου εργασία για την εδαφική ανάπτυξη τη πολιτική για τη συνοχή. Κύριο Βόν, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι και εγώ σύντομο στα σχόλιά μου, όπω και η προγραμματική Γιατί μα πιέζει ο χρόνο. Λοιπόν, καταρχήν, προ τον τίτλο τη έκθεση. Είναι πολύ σημαντική έκθεση, αλλά ο τίτλο ομολογώ ότι δεν είναι και πολύ συνεργαστικό. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι έχουν τα πράγματα, θα πρέπει να το αποδεχτούμε. Μην ξεχνάτε ότι σε αυτή τη φάση μιλούμε μόνο για έλλειμμα εργασία, αγαπητοί συνάδελφοι. Συνεχίζονται οι συζητήσει με την Επιτροπή, με του ενδιαφερομένου, συνεχίζονται οι διαβουλεύσει πριν αποκρισταλωθεί η μορφή τη έκθεση. Θα προτείνω εναρμόνιση των κανόνων και μεταξύ των ταμείων και ε, προταθούν συνέργειες μεταξύ των ταμείων. Βέβαια δεν ξέρουμε τι μηχανισμοί θα θεσπιστούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να υλοποιήσουμε το στόχο αυτό. Αυτόν. Πάντως ε, αυτό είναι το κενό που έχω εντοπίσει στον Γενικό Κανονισμό και νομίζω ότι το ανέφερε προηγουμένως και ο κύριος Βανίλστερόι. Η έκθεσή μου θα διερευνήσει πιθανούς μηχανισμούς για την ε, για τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των ταμείων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα σε κάποιες περιφέρειες και θα μιλήσω, θα προτείνω και με, μερικούς μελλοντικούς μηχανισμούς. Για παράδειγμα, μερικές περιφέρειες προτείνουν να δημιουργηθεί ένα ενιαίο πόρταλ, μια ενιαία θηρίδα για να μπορεί κανείς να υποβάλει έτσι για οποιαδήποτε από τα πέντε ταμεία. Επίσης έχουμε άλλα παραδείγματα Και αυτά τα παραδείγματα τα αναλύει η έκθεση. Επίσης εξετάζει τις προτάσεις του κανονισμού για να δούμε κατά πόσο στο μέλλον είναι χρήσιμοι παρόμοιοι μηχανισμοί. Πάντως, μερικές από τις προτάσεις της απλούστευσης, για παράδειγμα, θα τις χρησιμοποιήσουμε είναι χρήσιμες. Κίνη κανόνες, εφάπαξη, καταποκοπή ποσά, ηλεκτρονική συνοχή. Όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα ως προς την ε, συγκέντρωση των ταμείων, το συντονισμό των ταμείων και ο προσανατολισμός μας σε αποτελέσματα και όχι σε εκροές. Νομίζω αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό για καλύτερο συντονισμό των ταμείων. Επίσης, αναφέρεται και χρήση των χρηματοπιστωτικών ε, μηχανισμών. Και μάλιστα όσο προχωρεί ο καιρός, τόσο πιο σημαντικό θα είναι αυτό το θέμα για τα κοινωτικά ταμεία καλύτερο συντονισμό των ταμείων, χρησιμοποίηση νέων χρηματοπιστωτικών εργαλείων για συμπλήρωμα ε, κάποιων κονδυλίων. Νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καλύτερη απήχηση. Η έκθεση αναφέρονται και τα αστικά κέντρα, οι αστικές περιοχές. Ήδη το συζητήσαμε στην Επιτροπή πολλές φορές συμφωνούμε ότι οι πόλεις και οι αστικές ζώνες μπορούν να δημιουργήσουν κινητήριο μοχλό ανάπτυξης. Οι επενδύσεις πάντως στις ε, πόλεις και στα αστικά κέντρα από τα κοινοτικά ταμεία θα πρέπει να εξασφαλίσουν ε, απολαβή αυτών των κονδυλίων όχι μόνο από τις πόλεις, από το στερό περιβάλλον των πόλων, αλλά να, να ωφελούν την ευρύτερη περιοχή γύρω από τις πόλεις. Οπότε ο συνδυασμός των κονδυλίων θα πρέπει να εξασφαλίσει ε, την βελτίωση της κατάστασης όχι μόνο στις, ε, περιορισ... όχι μόνο στις πόλεις αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Σε ό,τι αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και αυτό είναι ε, θεμελιώδους σημασία. Αν θέλουμε πραγματικά καλύτερο συντονισμό των ταμείων ώστε να έχουμε καλύτερη απήχηση, καλύτερη αξιοποίηση των κονδύλιων. Αναφέρθηκαν κάποιες προτάσεις μηχανισμών. Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη με προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω σε τοπικό επίπεδο πρωτοβουλίες. Θα το στηρίξουμε γιατί με μια τέτοια προσέγγιση σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο θα έχουμε καλύτερη χρησιμότητα, καλύτερη ωφέλη, αλλά θα πρέπει να αποφύγουμε υπερβολικό γραφειοκρατικό άχθος. Αναφέρεται επίσης στην έκθεση τα κοινά σχέδια δράσης. Μπορούν έτσι να βελτιώσουν τη συνεργασία μεταξύ των περιφερειακών και τοπικών αρχών, αλλά και εδώ χρειαζόμαστε λεπτομεριακή ανάλυση των προτάσεων αυτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, ό,τι αφορά τις επενδύσεις εδαφικής συνοχής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα υπάρχοντα προγράμματα. Να χρησιμοποιήσουμε τις υποδομές και το δυναμικό που υπάρχει, να μην σπέβδουμε να δημιουργούμε νέα προγράμματα, να αξιοποιούμε τα υπάρχοντα. Αυτά είναι σημαντικό να συντονίσουμε τα ταμεία. Κρίμα που δεν μπορούμε σε ορισμένε περιπτώσει να συμπεριλάβουμε και τον ορίζοντα Ευρώπη 2000, γιατί θα μπορούσαμε εκεί να χρησιμοποιήσουμε τα ταμεία, αλλά έχουμε πολλούς στόχους να υλοποιήσουμε. Περιμένω και τα σχόλια των συναδέλφων. Θα έχουμε και δημόσια κρόαση με τους ενδιαφερομένους στο επόμενο δίμηνο και μετά από αυτό θα υποβάλω και το έγγραφο εργασία. Αυτή είναι η πρώτη ανταλλαγή υπόψη για αυτή την έκθεση ίδια πρωτοβουλία. Αν δεν κάνω λάθο, δύο είναι οι παρόντε και Σε Καλό χρόνο φίδου για να διεκπαιρεώσουμε τη συζήτηση σήμερα. Η κυρία Ουκατζεύσκα, πρώτη και συγητρία. Με ναι, δύο λόγια μόνο, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για το έγγραφο εργασία και την προθυμία του και τιμότητά του για συνεργασία προκειμένου να καταρτιστεί έκθεση. Πιστεύω ότι με αγαστή συνεργασία θα καταλήξουμε σε μια έκθεση που θα βελτιώσει την κατάσταση της περιφέρειας και θα τις βοηθήσει να λύσουν τα προβλήματά τους. Συμφωνώ με την πρόταση για την αστική διάσταση και συμφωνώ ότι θα πρέπει να καλύψουμε και θέματα του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και ζητήματα που αναφέρονται στο Γενικό Κανονισμό. Πάντως ε, ε, ήταν πολύ καρποφόρα και μέχρι τώρα συνεργασία και προσβλέπω σε συνέχιση και στο μέλλον μέχρι να διαμορφώσουμε την έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Χουισμένοβα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Θεωρώ ότι αποτελούν βήμα πρόοδου και επιτρέπουν τη χρηματοδότηση τοπικών στρατηγικών. Θα πρέπει ωστόσο να έχουμε υπόψη ότι για να προωθήσουμε αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να έχουμε ικανότητα και στον, ε, δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και στις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και επίσης χρειάζεται περισσότερο η πολιτική συνοχή ε, στις περιοχές εκείνες που ακριβώς, όπου ακριβώς λείπει. Ο κύριος Λαμ, ε, Φανίστηλροι. Πρέπει να πω ότι με παραξένεψε ο τίτλος. Μιλάει για ε, βελτιστοποίηση optimizing ή για αισιοδοξία optimism. Μήπως πρέπει να το ξαναδεί αυτό η Επιτροπή να εμπνευστεί από τον τίτλο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο και σημασία, νόημα αυτή το κείμενό σα, εάν ακολουθούσατε αυτό που είπε και ο κύριο Πίπερ, δηλαδή ότι χρειάζεται μια ολοκληρωμένη πολιτική, χρειάζεται μια πολιτική για τι τιμέ και μια προσέγγιση. Σε, με, με τα πέντε ταμεία. Είπατε τώρα εσείς ε, για την ε, περιφερειακή προσέγγιση και νομίζω ότι θα, ήταν καλό να κοιτάξουμε τι μπορούμε να ε, με, τι μπορούμε να επιφορτήσουμε τις δικές μας τις χώρες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν μιλάω μόνο για τα 82 ε, εκατομμύρια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή για την απασχολησιμότητα της νεολαίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε ε, συγκεκριμένες απαντήσεις, να βρούμε συγκεκριμένες απαντήσεις μέσα από την περιφερειακή μας πολιτική. Και άρα λοιπόν αντί να βελτιστοποιήσουμε την εδαφική ανάπτυξη με την ε, πολιτική συνοχής, θα πρέπει να προωθήσουμε τις ιδέες αυτές. Ε, μην ξεχνάτε ότι δεν προσφέρονται νέα μέσα και ίσως εάν αναδιαμορφώσετε το κείμενό σας μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Θέλετε να σχολιάσετε σύντομα κύριε Βόν. Πολύ σύντομα για τον Λάμπερτ. Ζητώ συγγνώμη για τον τίτλο τη εκθέσεως. Ίσως ήταν ε, κακή επιλογή. Ε, χαίρομαι που κάποιο τον βρήκε καλό. Μπες από μετά την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων, ίσως αντιληφθούν οι συνάδελφοι τι σημαίνει. Δύο σχόλια. Ένα για τι στρατηγικέ τοπική ανάπτυξη που θεωρώ ότι είναι πολύ καλέ και γι' αυτό είπα και εισαγωγικά ότι εάν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε αυτή την ηγετική θα έλεγα προσέγγιση θα πρέπει και οι μηχανισμοί που θα ε, εισαχθούν να μην είναι πολύ περίπλοκοι. Το είπατε και εσείς άλλωστε να μπορούν οι τοπικές κοινωνίες να αναπτύσσουν προγράμματα, σχέδια, έργα και να αξιοποιούν για αυτά διάφορα κονδύλια. Ο Λάμπερτ βλέπω ότι αναγνωρίζει δυναμικό στην έκθεση αυτή ε, δυνατότητες. Πιστεύω και το είπα και στην εισαγωγική μου παρατηρήση ότι τα κενά πάντοτε ήταν το πώς θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε τα ποσά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αλλά ε, πάνω απ' όλα νομίζω με τους εμπλεκόμενους φορείς, ε, αν τους πείθαμε και αν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε τη συνεργασία τους με παράλληλη άντληση από κοινού διαφορών ε, δυνατοτήτων χρηματοδότηση, θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε σημαντικά τις σε Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. βεβαίω. δεν έχει κλείσει η συζήτηση. Εν τω μεταξύ μπορείτε και να συνεργάζεστε ε, όσοι ενδιαφέρεστε. βεβαίω και οι, συγητές, οι Κλείνω τη συνεδρίαση. Έχουμε τώρα την ε, συνεδρίαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη μορφή τη ε, ομάδα εργασία για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ξανά συναντιόμαστε 29 Μαου Τρίτη και 30 Τετάρτη